Καλημέρα σας. Να σας υπενθυμίσω ότι αναμεταδίδεται η συνεδρίασή μας. Ε, εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, ε, θεωρούμε ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Σήμερα θα μας απασχολήσουν οι απειλές στον κυβερνοχώρο ο κύριος Γκρινμπερ και ο κύριος Κάρ, που ήταν, είναι οι υπεύθυνοι της μελέτης την οποία είχαμε ε, ζητήσει για την ε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. κυβερνοχώρο. Ο κύριος Βιλελόγκα επίσης ε, είναι εδώ για να μας ενημερώσει για την δουλειά που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προστατευτούμε από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Επίσης, Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ε, ε, πολύτιμη βοήθεια της ε, Κομισιόν. Οι απειλές στον κυβερνοχώρο είναι πολύ σημαντικές, είναι πολύ επικίνδυνες για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθεαυτή προσπαθεί, προσπαθούν να προστατευτούν από τις απειλές και από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Το ΝΑΤΟ το ίδιο κάνει μέσω από το κέντρο του στο Ταλίν. Επίσης, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, θεωρούν τις απειλές και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σαν πολεμικές επιθέσεις ε, τώρα το πρόβλημα ποιο είναι, ότι δεν μπορούμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τις επιθέσεις. Άρα η απάντηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μέχρι στιγμής στο ΝΑΤΟ έχει αποκλείσει το να θεωρηθούν ε, ε, πολεμικές ενέργειες οι επιθέσεις στον κυβέρνο χώρο. Όμως θέλει να προστατευτεί από τις επιθέσεις αυτές δημιουργώντας μια ειδική ομάδα έτσι ώστε να αντισταθούμε σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Θα δούμε εάν η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα μας δώσει κάποιες ε, ε, συμβουλές για το πώς θα μπορούσαμε να προστατευτούμε από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Καλό θα είναι να ακούσουμε τον κύριο Γκρίνμπαρκ και την κύρια την Μακλάρ που είναι και η υπεύθυνη για τη σύνταξη της ε, μελέτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ για την εισαγωγή. το όνομά μου είναι η Αλεξάνδρου Κλίνμπερκα, είμαι από το Ινστιτούτο διεθνούς πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε ξεκινήσει μία μελέτη για τις ε, επιθέσεις και για τις για τον πόλεμο αν θέλετε ε, στον κυβερνοχώρο ε, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι... Ε, υπάρχουν δύο τίτλοι στην μελέτη. Ε, το ένα αφορά τον κυβερνοχώρο και τις επιθέσεις και το άλλο μιλάει για τις εξουσίες, για τις δυνάμεις στον κυβερνοχώρο. Θα κάνω μια εισαγωγή μεν, αλλά αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να διαβάσετε την έκθεση αυτή καθεαυτή. Εγώ απλώς και μόνο θα αναφέρω ορισμένα βασικά σημεία Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να κάνουμε μια εισαγωγή ε, ούτως ή άλλως στον κυβερνοχώρο τα πάντα είναι αμφιλεγόμενα. Δεν υπάρχει και ούτως ή άλλως και η ίδια ορθογραφία. Cyber war στα αγγλικά είναι μία λέξη ή μπορεί να είναι δύο λέξεις. Υπάρχουν, υπάρχουν και υπάρχει, μπορεί να μπει και μία παύλα ανάμεσα. Αυτό μας δείχνει οι διαφορετικές ορθογραφίες ε, ε, δείχνουν και την, ε, τις διαφορές στην αντιμετώπιση. Δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες ανάμεσα ανάμεσα στα κράτη ε, δεν υπάρχει κοινός ε, ορισμός, ε, ο πόλεμος στον κυβερνοχώρο σημαίνει διαφορετικά πράγματα για άλλες χώρες. Υπάρχουν όμως και άλλες έννοιες που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο της πληροφορίας, με τις εξουσίες στον κυβερνοχώρο κτλ. Ούτε εκεί υπάρχουν ορισμοί. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν και ερωτήσεις που είναι, να είναι κοινέ. Τι ακριβώς θέλουμε να, να πετύχουμε, τι θέλουμε να εξετάσουμε. Επίσης, ποιες είναι οι ευαισθησίες Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι θα πρέπει να αναφερόμαστε ε, στον πόλεμο, στον κυβερνοχώρο με πολλού έντονους όρους. Άλλοι θεωρούν ότι αν μιλάμε έτσι ε, δημιουργούμε μια κάποια κλιμάκωση. Ε, πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι, εργάζομαι για το Αυστριακό Ινστιτούτο και είμαι επίσης και σύμβουλος της Αυστριακής Κυβέρνησης. Όμως εδώ αυτή τη στιγμή μιλάω σαν ένας απλός πολίτης και οι απόψεις μου δεσμεύουν μόνο τον ίδιο. Να σας δώσω κάποιες ε, βασικές ε, πληροφορίες όσον αφορά τις επιχειρήσεις ε, πληροφόρησης. Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε γιατί μιλάμε. Αυτό το οποίο θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι το Computer Network Operations που αποτελείται από τρεις βασικές μονάδες είναι οι επιθέσεις στο CNA, ε, στον, την εκμετάλλευση των δικτύων υπολογιστών, το, ε, ε, η κατασκοπία και το CND που είναι η άμυνα. Οι επιθέσεις όμως στα δίκτυα των υπολογιστών είναι ένας ορισμός. Επομένως για να γίνει μια τέτοια επίθεση πρέπει να έχουμε και εκμετάλλευση και επίθεση. Θα πρέπει να, τα δούμε, να τις δούμε όλες, όλες τις ε, διαστάσεις ε, του προβλήματος. Ε, δεν ξέρω αν φαίνονται εδώ στις διαφάνειες. Έχουμε διάφορα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Τώρα, θα ήθελα να μιλήσω λίγο περισσότερο για το cyber power, για την δύναμη, για την εξουσία του στον κυβερνοχώρο. Ε, ο πόλεμος ε, του κυβερνοχώρου, στον κυβερνοχώρο, το cyber warfare, ε, είναι μια μεταφορά αν θέλετε και μια άλλη μεταφορά είναι το cyber power. Cyber power τι είναι, είναι στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται, μπορεί και, στο, και να περιλαμβάνονται στο cyber warfare, αλλά όχι εξαντλητικά. Έχουμε συνεργασία, επίθεση, ε, και έχουμε τον, ε, και τα, τις υπηρεσίες υποστήριξης αν θέλετε ε, για την τρομοκρατία και για τις τρομοκρατικές ενέργειες. Το βασικό θέμα ποιο είναι, ότι το cyber power, η δύναμη, η εξουσία αν θέλετε, συμπεριλαμβάνει ένα σωρό στοιχεία ναι, όντω μιλάω πάρα πολύ γρήγορα, ζητώ συγγνώμη και ζητώ συγγνώμη και του Λοιπόν, το Cyber Power ε, εκπροσωπεί διάφορες εντολές αν θέλετε και όσον αφορά την, ε, τον πόλεμο πληροφόρησης και όσον αφορά το Cyber Warfare. Όταν μιλάμε για warfare, για πόλεμο, όντως ε, μιλάμε και για στρατιωτική διάσταση αν θέλετε. Λοιπόν, εδώ έχουμε την διακυβέρνηση του κυβερνοχώρου, έχουμε τις επικοινωνίες, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, στην προστασία των υποδομών, ε, τις συγκρούσεις, αν θέλετε, ε, πώς, ρυθμίζονται οι συγκρούσεις, η σύμβαση της Γενέβης, παραδείγματος χάρη, και η τρομοκρατία. Υπάρχουν πολλές εντολές, αν θέλετε, πολλές, πολλά στοιχεία που ε, συμπεριλαμβάνονται στο cyber power, που δεν είναι μόνο cyber warfare, είναι θέματα της αστυνομίας, των ε, Υπουργείων Άμυνας ε, ε, και άλλων εξουσιών, αν θέλετε, πέραν του, των στρατιωτικών. Τώρα, όπως σας είπα, ένα βασικό πρόβλημα σε όλες τις σε όλα τα προβλήματα εδώ στον κυβερνοχώρο είναι να εντοπίσουμε τον υπεύθυνο δεν μπορούμε να δούμε ποιο είναι υπεύθυνο για την επίθεση στον κυβερνοχώρο. Αυτό μπορούμε να το δούμε εκ των υστέρων. Αλλά ε, στη στιγμή που διαδραματίζεται δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Καταρχάς δεν μπορείς να ξέρει αν είναι μια, ένα έγκλημα, μια τρομοκρατική ενέργεια ή μια πολεμική μια επίθεση. Διότι η εκμετάλλευση των δικτύων ε, υπολογιστών είναι ένα, αν θέλετε, μια, μια προϋπόθεση για μια επίθεση σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Μπορεί να σας πούν ότι η κατασκοπία αυτή δεν είναι ένα θέμα ασφάλειας. Μπορεί να μην είναι θέμα ασφάλειας αυτό ο καθεαυτό. Αλλά τα ίδια κανάλια που χρησιμοποιούνται για την κατασκοπία ε, για, το, για τους υπολογιστές μπορούν να οδηγήσουν, να μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ε, άλλες επιθέσεις. Είναι δηλαδή ένα βήμα. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να τονίσω είναι ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στα θέματα του, του εγκλήματος ή της τρομοκρατίας. Το ένα είναι η αντίσταση και το άλλο είναι η αποθάρρυνση. Δηλαδή καταρχάς το ένα είναι το πρώτο η αντοχή και η αντίσταση είναι να μην γίνει, να, να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την επίθεση και η αποτροπή αν θέλετε είναι να περιορίσουμε τις ζημιές. Αυτό θα πρέπει να πούμε είναι ε, ότι εδώ γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για αυτές τις δύο αρχές αν θέλετε, οι, κυρίως στις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα επανέλθουμε στις ΗΠΑ σε λίγο, αλλά και στην Ευρώπη ε, ασχοληθήκαμε πολύ με την αντοχή ή την αντίσταση και λιγότερο με την αποτροπή. Βέβαια, δεν μπορείς να έχεις μία μια πολιτική που να είναι 100% ε, στηριγμένη στην αποτροπή ή 100% ε, να στηρίζεται στην αντίσταση, χρειάζεται να κάνουμε ένα μείγμα. Εμείς θεωρούμε ότι η αντίσταση ή η αντοχή είναι καλύτερο. Ε, βέβαια χρειάζεται και, και κάποια στοιχεία αποτροπής. Ας δούμε τώρα ποιες είναι οι βασικές ε, εξουσίες ε, στον κυβερνοχώρο. Οι Κινέζοι στηρίζονται κυρίως στην αντίσταση, στην αντοχή. Στο στρατιωτικό τομέα προσπαθούν να προστατεύσουν κυρίως τον κυβερνοχώρο τους Υπάρχουν όμως βασικές αλλαγές ανάμεσα σε αυτά τα οποία ε, κάνουν ε, στις, οι εθνοφύλακες, ε, οι παραστρατιωτικές οργανώσεις, οι, οι, συγγνώμη, εφεδρίες τους ή το Υπουργείο Άμυνας. Οι Κινέζοι θέλουν να διατηρήσουν και να προστατεύσουν τα συστήματα ε, πληροφορικής τους. Έχουν ένα δικό του σύστημα, το Coolen. Έχουν τα δικά τους microchips, τα οποία δεν μπορούν να μολυνθούν αν θέλετε, αλλά και έχουν και άλλους μηχανισμούς άμυνες. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν ε, προγράμματα λογοκρισίας, πολύ αυστηρά προγράμματα λογοκρισίας. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μέρος των δυνάμεων ασφάλειας θέλουν να προστατεύσουν τις εσωτερικές δραστηριότητες στην Κίνα αλλά και εκτός Κίνας. Βέβαια το πρόβλημα είναι και πώς ε, γίνονται οι ορισμοί, ποιους ορισμούς χρησιμοποιούμε. Πριν από μερικές εβδομάδες οι Κινέζοι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, έχουν 450 εκατομμύρια χρήστες του ίντερνετ και από αυτούς ε, υπάρχουν 200 εκατομμύρια blogs ε, και με τον έχετε με τον τρόπο αυτό μια ιδέα για το πόσο ε, δονείται αν θέλετε ο κυβερνοχώρος στην, στην Κίνα και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ανησυχεί, ανησυχεί ιδιαίτερα για τον κυβερνοχώρο δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι οι αρχές στην Κίνα προσπαθούν να προστατευτούν, αν θέλετε, να ελέγχουν αυτούς τους ε, χρήστες ε, του, του ίντερνετ για να μπορούν να ε, συνεργάζονται, αν θέλετε, με τους netizens σε σχέση με το citizens που είναι μια, ένας όρος που εφήβρανε οι Κινέζοι. Μπορώ να σα μιλάω για τα θέματα αυτά για ώρα και εδώ μου ζητάνε να τα πω σε δύο λεπτά, αλλά τέλο πάντων για να συνοψίσω. Οι περισσότερε ικανοστρατιωτικέ κανότητε τη Κίνας είναι αμυντικέ και ε, προσπαθούν να προστατευτούν και από τις επιθέσεις από το εξωτερικό και κυρίως από τις ΗΠΑ, αλλά πιο σημαντικό να αμήνονται από επιθέσει που θα προέρχονται από το εσωτερικό τη χώρα. Ε, προσπαθούν να προστατευτούν από τους Κινέζους hackers αλλά και θέλουν να κρατήσουν αυτούς τους hackers ε, απασχολημένους. Δηλαδή προσπαθούν να ε, στρέψουν τους Κινέζους αυτούς hackers σε επιθέσεις εναντίον των Αμερικανικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τους λένε σταθείτε εκεί και όχι σε εμά. Τώρα για τους Ρώσους. Είναι soft deterrence έχουν χαρακτηριστεί οι ικανότητες της Ρωσίας. Ποιο είναι το πρόβλημα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να ελέγχεται η... Uh, Russia, for instance, has probably the unique ability. Ε, ε, ελέγχουν τα πάντα η, η υπηρεσία ασφάλειας ε, της, της Ρωσίας. Δεν υπάρχουν πολλές χώρες που μπορούν να το κάνουν αυτό. Ε, και υπάρχει και έχει οθετηθεί και η κατάλληλη νομοθεσία. Κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το κυβερνοέγκλημα στην Ρωσία ε, είναι το αποτέλεσμα του, της, του προηγμένου εκπαιδευτικού συστήματος της Ρωσίας. Είναι πάρα πολύ προηγμένη. Το 40% του ε, κυβερνοεγκλήματος την προηγούμενη χρονιά οφείλεται στους Ρώσους. Οι ε, υπεύθυνοι είναι οι, είναι υπεύθυνες ρωσικές εγκληματικές ομάδες. Υπάρχουν και άλλε εγκληματικέ ομάδες οι οποίες δρούν από το ρωσικό έδαφος, αλλά και η, η ρωσική εγκληματικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχουν ε, πολλές... Ε, το δεκαετία του 1990 και στις αρχές δεκαετία του 2000 ε, υπήρχε και, υπήρχαν και διάφορες υποψίες για σχέσεις ανάμεσα στις υπηρεσίες ασφάλειας και στο οργανωμένο έγκλημα. Και Υπάρχουν κάποια σημεία πίεση, όπω παραδείγματο χάρη οι πατριώτε hackers, που είναι εθνικιστές, τους οποίους χρησιμοποιούν και οι και οι αρχές ε, παραδείγματος χάρη για να οργανώσουν επιθέσεις στη Γεωργία, στην Τσετσενία ε, και με την υποστήριξη κάποιων ομάδων νέων που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να επιτεθούν στους εξωτερικούς εχθρούς αλλά και στους εσωτερικούς. Αναφέρθηκα στις ρωσικές ικανότητες σαν soft deterrence. Ε, το πιο σημαντική, γιατί το πιο σημαντικό ε, κομμάτι ε, για τους Ρώσους δεν είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε, είναι αυτό το οποίο δεν γνωρίζουμε. Τώρα, στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, είναι ακριβώς το αντίθετο. Και βλέπετε εδώ σε αυτόν τον κατάλογο ποιος, πόσες οργανώσεις εμπλέκονται στην προστασία του κυβερνοχώρου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δαπανούν τεράστια ποσά, πολύ περισσότερα από όλοι ο υπόλοιπος κόσμος μαζί. Ε, οι επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο είναι κυρίως στρατιωτικές, είναι επιχειρήσεις, επιχειρησιακές ε, δραστηριότητες. Ε, δεν τους ενδιαφέρουν να σβήσουν τα φώτα, αλλά να σβήσουν τα συστήματα ραντάρ και είναι, έχουν ένα αμυντικό χαρακτήρα. Λόγω ακριβώς του μεγέθους των Ηνωμένων Πολιτειών πάρα πολλά χρήματα ε, θέλουν να, να ε, δίνονται για να ε, προστατεύσουν το δίκτυο πληροφοριών Βέβαια, έχοντα δώσει όλα αυτά τα χρήματα ε, και έχοντα όλε αυτές τι οργανώσει. όλες αυτές τις οργανώσεις, το θέμα της αντίστασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το πρόβλημα είναι το μέγεθος, επίσης άλλο πρόβλημα είναι η ευελιξία. Το μέγεθος των Ηνωμένες Πολιτείε είχαν ε, ε, στηριχθεί κυρίως στην αποθάρρυνση, στην αποτροπή. Είναι γιατί λέγανε ότι οποιασδήποτε επιθέσεις και αν γινόντουσαν και όσο κακό για κάνανε αυτές επιθέσεις, εμείς έχουμε έχουμε τα μέσα και τα τεχνολογικά αλλά και τα οικονομικά για να το ξεπεράσουμε. Αυτό ήταν η αρχή που ακολούθησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε εδώ και χρόνια. Είχαμε και την πυρηνική αποτροπή. Ε, τώρα πώ μπορεί να λειτουργήσει αυτό σε περίπτωση που θα υπάρχουν τρομοκρατικέ επιθέσει στον κυβερνοχώρο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί δεν μπορούμε να, το, να αντισταθούν. Ε, και επίση το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποιο είναι αυτό ο οποίο επιτίθεται στον κυβερνοχώρο. Τώρα, το πρόβλημα δεν είναι επίση πώς θα προστατεύσουμε την, ε, τις κρίσιμες υποδομές, αλλά ότι μπορεί να υπάρχουν ε, και επιθέσεις στην, ε, βιομηχανική, στην βιομηχανία των Πολιτειών. Βέβαια, όλες αυτές, όλες αυτές οι οργανώσεις δεν λειτουργούν στα πλαίσια των κυβερνητικών της, της κυβέρνησης, είναι εκτός κυβέρνησης. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην συνάδελφό μου η οποία θα μιλήσει για την διακυβέρνηση στο ίντερνετ και για τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες. Καλημέρα και από μένα, είμαι η Χάιντε Μακλάρθ, εγώ θα σας μιλήσω Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι εκπροσωπώ το Εστονικό Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών, άρα εκφράζω καθημαϊκές απόψεις ως επιτοπλίστων που σε ανταπο... αντικατοπτρίζουν τις επίσημες αστυνομικές θέσεις, τις θέσεις της αστυνομικής κυβέρνησης δηλαδή. Μιλάμε λοιπόν για την ασφάλεια, για τον πόλεμο και για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι περισσότερες κυβερνοδραστηριότητες διεξάγονται όχι στον κρατικό τομέα αλλά στον ιδιωτικό τομέα. Το 80% των κρατικών ε, υποδομών, των κρίσιμων υποδομών βασίζονται στον ηλεκτρισμό, στο νερό, στις μεταφορές. Χρησιμοποιούν συστήματα πληροφοριών, κυβερνοσυστήματα. Και ε, αυτό το τεράστιο τμήμα της κοινωνίας μας αποκαλείται κρίσιμη υποδομή, κρίσιμες υποδομές που στηρίζονται από τα συστήματα πληροφοριών. Η ομαλή ε, λειτουργία αυτών των συστημάτων πληροφοριών αποτελεί τον πυρήνα του μη στρατιωτικού ε, σκέλους της κυβερνοασφάλειας. Και μετά από την επεξήγηση αυτή θα σας μιλήσω για κάποιες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται μέσα στον κυβερνοχώρο χώρο. Νομίζω ότι ο Αλεξάνδρ παρουσίασε πληρέστατα τις διάφορες δυνατότητε των μεγάλων κυβερνοδιάμενων, ιδίω από την στρατιωτική ε, διάσταση. Εγώ θα περάσω στην ε, πολιτική, τη μη στρατιωτική διάσταση της κυβερνοασφάλειας και θα σας ε, αναφέρω πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μέχρι σήμερα. Πρώτα απ' όλα, Έχουμε την ε, διακυβέρνηση του διαδικτύου, το Internet Governance. Το διαδίκτυο, ε, όταν ε, πρωτοδημιουργήθηκε, πριν από τρεις δεκαετίες περίπου, δεν είχε αυτές τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική υποδομή. Όλα τα κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθούν να βρουν λύσεις για να υπάρχει ένα διαφανές καλό μοντέλο διαδικτυακής διακυβέρνησης, η οποία μέχρι σήμερα γίνεται στον τομέα, τον τεχνικό στον τομέα της πολιτικής. Και είναι μια διαδικασία από κάτω προς τα πάνω, bottom-up. Έχουμε τους ε, μηχανικούς του διαδικτύου, οι οποίοι προσπαθούν να προσδιορίσουν τις τεχνικές δυνατότητες ε, του διαδικτύου. Το έχουν καταφέρει πολύ καλά μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Στον τομέα της πολιτικής έχουμε κάποιους φορείς όπως είναι η ICON που είναι η εταιρεία για την απόδοση αριθμών και ονομασιών του διαδικτύου. Έχουμε και την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Βέβαια συχνά κατηγορείται ότι η πρώτη, ε, η ICON δεν έχει πάρα πολύ διαφανή ε, λειτουργία. Επί της ουσίας, στην ε, διαδικτυακή διακυβέρνηση δύο σημαντικά ζητήματα υπάρχουν. Το θέμα της ελευθερίας του διαδικτύου αφενός και το θέμα της διαδικτυακής ασφάλειας αφετέρου. Οι δημοκρατικές χώρες δεν έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία να αλλάξουν το τρέχον μοντέλο, το οποίο είναι πολύ ε, κλαδικό, έχει πολυμερές θα έλεγα. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες, πολύ ενδιαφερόμενοι φορείς Κάποιε κυβερνήσει θα ήθελαν ο ρόλο ε, ο κρατικό να είναι μεγαλύτερο στη διαδικτυακή διακυβέρνηση και φυσικά υπάρχουν και κάποιες χώρες που δεν είναι τόσο δημοκρατικές που ε, θέλουν να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο και υπάρχουν και κάποιες οργανώσεις που ενδιαφέρονται να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στη διαδικτυακή διακυβέρνηση. Μέχρι στιγμής πάντως ε, δεν φαίνεται να υπάρχει συνένεση για το βασικό μοντέλο ένα core model και το multi ε, stakeholder model, αυτό που ισχύει δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει πολιτική και οικονομική επιρροή, είναι ένας παγκόσμιος ε, παράγων, θα μπορούσε ίσως να εκφράσει μια σαφή άποψη και να διατυπώσει καλύτερες προτάσεις για την διαδικτυακή διακυβέρνηση και σε σχέση βέβαια με τη συνεργασία που θα μπορούσε να υπάρχει με τις ΕΙΠΑ για την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου εφόσον βέβαια βρεθεί ένα τέτοιο νέο μοντέλο. Αυτό βέβαια εντάσσεται στι ε, υποδείξει. Απλά ακολουθώντα τη συλλογιστική μου, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει σε αυτό το πλαίσιο. Έχουν επίση αναλυφθεί κάποιε παγκόσμιε πρωτοβουλίε Υπάρχει δραστηριότητα, μεν, αλλά δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχουμε την κοινότητα της κυβερνοασφάλειας που προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να αυτορυθμίσει τον τομέα της πολιτικής. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές ανεπίσημες πληροφορίες. Στο Meridian Forum πρώτα απ' όλα, όπου έχουμε κάποιους ε, χαράκτε πολιτική οι οποίοι ανταλλάσσουν ε, τις βέλτιστες πρακτικές σε, ε, σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουμε και το Forum που first, δηλαδή για την ανταπόκριση, την αντίδραση σε κάποια συμβάντα, και την ασφάλεια. Έχουμε ομάδες εμπειρογνωμόνων και από τον κρατικό τομέα και από τον ιδιωτικό τομέα που ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και όντας εστονή το 2007 νομίζω ότι μας έσωσαν αυτά τα φόρουμ τα ανεπίσημα και όχι τόσο η κρατική δράση, η δράση της κυβέρνησης γιατί αυτά τα ανεπίσημα δίκτυα που λειτουργούν σε όλες τις ε, χώρες μεταξύ ειδικών στον τομέα της ασφάλειας και από τη χώρα μας και από άλλες χώρες είχαν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και ανταπόκριση και έτσι μπορέσαμε και εμείς να προστατευτούμε από την επίθεση που είχαμε δεχθεί τότε. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες πρωτοβουλίες από πολυμερείς οργανισμούς. Πρώτα απ' όλα ένα πάρα πολύ σημαντικό νομικό εργαλείο που είναι η Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ίσως το μόνο νομικό μέσο που ε, θέτει κάποια πρότυπα για την ε, νομοθεσία των κρατών μελών. Επίσης, απαιτεί την συνεργασία για την επιβολή της νομοθεσίας μεταξύ των συμβαλωμένων. Οι περισσότερες χώρες ε, το έχουν, ε, έχουν επικυρώσει τη σύμβαση αυτή, όχι όλες. Οι ΕΠΑ έχει, ε, υπέγραψαν όπως και η Ιαπωνία και ο Καναδάς και άλλοι και επικυρώσει αυτή τη σύμβαση. Οι προηγμένες δηλαδή οικονομίες των χωρών όσα γενικότερα έχουν υπογράψει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης προωθεί αυτό το, το νομικό μέσο γιατί έχει να κάνει με πολύ σημαντικά ζητήματα που, αφορούν τον κυβερνοχώρο, το κυβερνοέγκλημα και την επιβολή της εσωτερικής νομοθεσίας. Και ίσως ε, να, μην χρειάζεται κάποιο άλλο νομικό μέσο. Μετά έχουμε την ομάδα εργασίας ε, του ΟΣΑ για την ασφάλεια των πληροφοριών και την, ε, τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα. Ο έχει επίσης διατυπώσει πολύ καλές συστάσεις ε, για την προστασία των κρίσιμων υποδομών. Είναι μια λέσχη πλούσιων χωρών βέβαια και απαιτεί από τα κράτη-μέλη του να έχουν ένα κατώτατο επίπεδο προστασίας ε, των ε, κυβερνοϊποδομών από οργανωτικής και τεχνολογικής πλευράς. Έχουμε στη συνέχεια τον ΟΑΣΕ για την συνεργασία και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Πολιτικο-στρατιωτική διάσταση της κυβερνοασφάλειας περισσότερο. Και έχουν ξεκινήσει εκεί να συζητούν ε, τα πρότυπα κρατικής ε, συμπεριφοράς. Φέτος μάλιστα αποφάσισαν ε, στον ΟΑΣΕ να συνεχίσουν με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης για τα κράτη εντό του κυβερνοχώρου με στόχο να μειωθούν οι κίνδυνοι παγκόσμιων ε, εσφαλμένων υπολογισμών και θέλουν να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια μεταξύ κρατών. Επί παραδείγματι, Εάν δείτε να έρχεται, είσαστε στο, στη διοίκηση στη, του κυβερνοχώρου στη ΣΥΠΑ και βλέπετε να έρχεται μια πολύ μεγάλη επίθεση από τη Ρωσία. Θα πρέπει να ξέρετε αν Πρόκειται για μια επισήμως εχθρική στάση ε, ή δράση από την κυβέρνηση της Ρωσίας ή ας πούμε της Κίνας ή αν κάποιος μη κρατικός φορέας ε, εξαπατά κατά κάποιο τρόπο, παραπλανεί και σας κάνει να πιστεύετε ότι προέρχεται η επίθεση από μια συγκεκριμένη χώρα. Για να επαληθευτεί λοιπόν ο, ε, μάλλον η προέλευση θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προθέσει τη χώρα. Είναι λίγο η ψυχροπολεμική λογική ουσιαστικά, σαν αυτά που γίνονταν μεταξύ Ρωσίας και ΕΙΠΑ. Με το πυρηνικό όπλο. Κανείς δεν ξέρει αν ήταν λάθος ή αν ήταν μια σκόπιμη κίνηση. Αυτή η λογική λοιπόν υπάρχει και στις ε, κυβερνοσυγκρούσεις. Επίσης, περνάμε τώρα στα Ηνωμένα Έθνη και τις δραστηριότητες τους, στον τομέα της πολιτικής, ε, πολλές πολιτικές και πολλοί τομείς δεν θέλω να σας επαναλάβω ή να αναφερθώ συγκεκριμένα ε, στον καθένα τομέα, αλλά έχουν ε, ψηφιστεί σημαντικά ψηφίσματα σε επίπεδο ΙΕ, τα οποία τονίζουν την κουλτούρα, αν θέλετε, της κυβερνοασφάλειας, το θέμα της ε, πρόληψης, το θέμα της αντοχής, της ανθεκτικότητας. Το 2009 στην Επιτροπή Αφοπλισμού ελήφθη μια σημαντική απόφαση, ψηφίστηκε ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα που αποφασίζει ότι θα εκπονηθεί έκθεση από τον ΟΗΕ για την κυβερνοασφάλεια στο πλαίσιο της εσωτερικής ασφάλειας. Η έκθεση αυτή έκθεση ε, η οποία εκδόθηκε το 2010 και είναι γνωστή ως η έκθεση της ομάδας κρατικών εμπειρογνωμόνων ε, έχει εξετάσει τα εξής θέματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν νόμοι που θα ισχύουν στον χώρο αν έχουμε μια σύγκρουση αντιπαράθεση μεταξύ χωρών. Ναι, λέει αυτή η έκθεση. Ε, σύγκρουση ενόπλων δυνάμεων, παραδείγματο χάρη. διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτά ισχύουν σε περίπτωση και ε, κάποια σύγκρουση στον κυβερνοχώρο. Μια ε, ένα άλλο συμπέρασμα αυτής της έκθεσης είναι ότι οι χώρες πρέπει να συνεργάζονται και να οικοδομούν μηχανισμούς ε, για την, πρόορη, για την έγκαιρη προειδοποίηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων και επίσης υπάρχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας για μια χώρα η οποία επιτεθεί με δεχθεί επίθεση μέσω ε, μέσων. Έχει το δικαίωμα αυτό άμυνα χώρα που δέχεται επίθεση. Και σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης αναφέρεται ρητά ότι αυτό ισχύει για τις χώρες. Από το ίδιο πάντα πλαίσιο, το πιο πολύ στρατιωτικό, ας δούμε τι κάνει το ΝΑΤΟ. Μετά το 2007, ε, οπότε και κατελήφθη ξαπίνη στο ΝΑΤΟ με την επίθεση αυτή που δέχτηκε η Εστονία, άρχισε να ασχολείται περισσότερο με το θέμα αυτό. Υπάρχει ε, το Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση των Κυβερνοεπιθέσεων, το οποίο συγκροτήθηκε στο ΝΑΤΟ. Είχε βέβαια ήδη κάποιε τεχνικέ δυνατότητες στο ΝΑΤΟ, ε, που είχε να κάνει πιο πολύ με την ανταπόκριση του ΝΑΤΟ σε κάποια συμβάντα στον κυβερνοχώρο. Έχουμε το, τη στρατηγική, ε, το στρατηγικό κόνσεπτ, το στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ, ε, το οποίο ε, διατυπώθηκε το 2010 και που λέει ότι το ΝΑΤΟ ε, θα μπορεί να αντιδράσει κατά οποιασδήποτε απειλής μεταξύ αυτών και κύβερνο απειλών και βέβαια των αναδυόμενων προκλήσεων στο τομέα της ασφάλειας. Και το 2011 το ΝΑΤΟ επικαιροποίησε την πολιτική για την κυβερνοάμυνα και ένα πρόγραμμα δράσης που υιοθέτησε με τρεις κατηγορίες απάντησης ή ανταπόκρισης από το ΝΑΤΟ. Πρώτη, συλλογική απάντηση σε μια τέτοια κυβερνοεπίθεση μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, επίθεση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σύγκρουσης ή ως μέρους, ως τμήματος συμβατικού πολέμου το σύστημα και οι διεργασίες για τη διαχείριση αυτής της ανταπάντησης. Δεύτερη κατηγορία απάντησης από το ΝΑΤΟ θα είναι αν η σύμμαχη ή ένα σύμμαχος θα είναι αντικείμενο κυβερνοεπίθεσης. Θα υπάρχει συντονισμένη απάντηση, ανταπάντηση από το ΝΑΤΟ. Και τρίτη κατηγορία θα είναι με τα ίδια δίκτυα του ΝΑΤΟ, αν αυτά τα ίδια δίκτυα υποστούν επίθεση, θα υπάρξει ανταπάντηση αμέσως από το ΝΑΤΟ ως Τώρα, μετά από αυτό ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Τι κάνει και τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε αξιόλογες δραστηριότητες υπό το πρίσμα της πολιτικής της ε, για την κυβερνοασφάλεια πολιτικού επίπεδου μέτρα. Πολλές πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν από την αρχή του 2000, της δεκαετίες του 2000. Ίσως η πρώτη πραγματική κυβερνό ας το πω, κυβερνοπρωτοβουλία που ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Ένωση να κινητοποιηθεί ήταν η οδηγία του 2005 του Συμβουλίου για τέτοια κυβερνο ε, ε, θέματα ε, επιθέσεων. Είχαμε και κάποιες δραστηριότητες από πλευράς κυβερνοτρομοκρατών και το 2009 ή 2010 πιθανότατα ήταν τα πιο σημαντικά χρόνια έτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πρωτοβουλίες ε, για την, αντιπολέμ... για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και τώρα υπάρχει μια πολύ σημαντική οδηγία για τα... την αντιμετώπιση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν θα έλεγα πιο, λειτουργικές, ε, ε, πιο λειτουργικά πλαίσια για την ε, δρομολόγηση αυτών των πρωτοβουλειών το κέντρο για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος το 2013 θα αρχίσει να λειτουργεί όπως ακούσαμε και από την Επίτροπο Μάνστρομ Τούτων λεχθέντων λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τις δραστηριότητες για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος και των συναφών δραστηριοτήτων διότι οι περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις μέχρι σήμερα στρέφονται στις οικονομικές, ε, στους οικονομικούς οργανισμούς ε, και θεσμικά όργανα και για ε, οικονομικά συμφέροντα υπάρχει απώλεια μεγάλων όγκων χρηματικών και η αρχές επιβολής του νόμου η αστυνομία δεν, επαρκεί να, δεν επαρκούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις επιθέσεις. Ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο που στρέφονται κατά των συμφερόντων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και εταιριών. Αυτό είναι ένα από τα δυνατά σημεία που έχει σαφώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί σε διεθνικό, διεθνές επίπεδο να δρομολογήσει πρωτοβουλίες και να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι περισσότερο για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Ένα άλλο σημαντικός πυλώνας για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος είναι η προστασία των κέριων υποδομών. Και βλέπουμε εδώ και στον πολιτικό τομέα ότι έχει κύρια σημασία δεν είναι μόνο η πρόληψη και η διασφάλιση έναντι εγκλήματος και όπως ε, ανέφερα και στην αρχή όλοι εξαρτώμαστε από τις ε, υποδομές αυτές. Καθημερινά οι κοινωνίες μας ε, εξαρτώνται όλο και περισσότερο από αυτά τα πληροφοριακά συστήματα δεν το αντιλαμβάνεται κανείς μέχρι ότου να συμβεί κάτι που δεν πάει καλά και να ε, σημειωθεί ένα πλήγμα. Όμως για αυτούς όλους τους λόγους οι κύριες ε, πρωτοβουλίες για την προστασία των υποδομών και η οδηγία για την Critical Infrastructure, Infrastructure Protection του 2008 είναι πολύ σημαντικά θέματα. Έχουμε και τον κατάλογο των υποδομών και της προστασίας τους διασύνοριακά. Ελπίζουμε ότι ο τομέας ε, για την προστασία αυτών των υποδομών θα λαμβάνεται όλο και περισσότερο υπόψη. Είδαμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και πριν από το 2007 και τα συστήματα για την περισσότερο ασφαλή πληροφορία και πληροφόρηση. Το 2009 είχαμε την ανακοίνωση προστασία της Ευρώπης από μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις και ε, παρεμβολές, διευρύνοντας ε, την ετοιμότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Και βλέπουμε ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό έτος ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε να προβληματίζεται πιο σοβαρά για αυτά τα θέματα και υπήρξε και ευρύτερη ε, κινητοποίηση. Το 2009 είχαμε μια ισχυρή οδηγία που υπερβλήθη το, η οδηγία πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες όπου πολλές οδηγίες παλαιότερες συγχωνεύθηκαν σε αυτό το ενιαίο πλαίσιο. Υπάρχουν ισχυρές συστάσεις για εταιρείε ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναφέρουν αμέσως περιπτώσεις ε, ε, δεδομένα τέτοιων κυβερνοεπιθέσεων ώστε να μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να τα αντιμετωπίσουμε. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις Υπηρεσίες Ασφάλειας όπου διοργανώθηκε από πλευράς του το πρώτο κυβερνο, η πρώτη άσκηση αντιμετώπισης ε, κυβερνοεπιθέσεων. Στο πολιτικό επίπεδο κινούμαστε προς την ορθή κατεύθυνση με τους ορθούς προσανατολισμούς. Ε, αξιόλογες πρωτοβουλίες ε, δρομολογούνται και θα πρέπει εδώ να υπάρξει ίσως ένας πιο έντονος συντονισμός, ο συντονισμός μεταξύ των πολιτικών αυτών πρωτοβουλειών που είναι αναγκαίο στοιχείο. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Και τώρα περνάμε στην κοινή πολιτική ασφάλειας ε, από πλευρά τη Ευρώπης. Μέσα σε αυτό το περιθώριο υπάρχει ακόμα πλαίσιο για βελτιώσεις. Ε. Η κυβερνοασφάλεια αναφέρθηκε στην έκθεση της υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ασφάλεια. Και υπήρξαν και πιέσεις που ασκήθηκαν ώστε να μπορέσει αυτή η πτυχή να ενταχθεί στην έκθεση. Υπάρχουν και πρακτικές πρωτοβουλίες, πιο χειροπιαστές πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και πιο πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Διπλωματική Υπηρεσία εξέδωσε, δρομολόγησε κάποιες καλές συστάσεις που δεν αντανακλώνται όμω στην έκθεση διότι είναι τόσο πρόσφατες. Μετά στη συνέχεια είχαμε και περισσότερο πληροφοριακά θέματα, ενημερωτικά θέματα Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία υποσυζήτηση μετά τις ε, τελευταίες ε, επιθέσεις που είχαν υποστεί τα θεσμικά όργανα. Είναι η σωστή συγκυρία χρονικά, το σωστό πλαίσιο να γίνουν όλα αυτά. Μα ζητήθηκε να συζητήσουμε την ετοιμότητα των κρατών μελών στην έκθεσή μας και να δούμε τι γίνεται με αυτήν. Κάναμε μια επισκόπηση σε σχέση με το έργο αυτό. Ουσιαστικά το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία ήταν αυτές οι τρεις μεγαλύτερες χώρες που μας απασχόλησαν που έχουν δρομολογήσει εσωτερικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος και για την κυβερνοασφάλεια και έχουν δρομολογήσει τέτοιες δράσεις με συγκεκριμένες δομές και κάποιες μεσαίων διαστάσεων, ενδιάμεσες, ε, ενδιάμεσων διαστάσεων χώρες έχουν και αυτές δραστηριοποιηθεί όσον αφορά τον ε, εθνικό μηχανισμό αντιμετώπισης ε, κυβερνοεπιθέσεων και διασφάλισης κυβερνοασφάλειας. Καθώς αυτό είναι κάτι το καινούριο, πολλές χώρες προβληματίζονται και σκέπτονται να δουν τι μπορούν να κάνουν και ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια περισσότερες χώρες θα συμμετάσχουν και θα δρομολογήσουν τέτοιες στρατηγικές για την προστασία του κυβερνοχώρου και θα επενδύσουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Για συστάσεις και συμπεράσματα λοιπόν θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Αλέξανδρο και πάλι. Παρακαλώ Αλέξανδρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι θα δούμε ένα προς ένα τα θέματα πυρήνα της μελέτης μας ε, για να κάνουμε κάποιες αξιολογήσεις και συστάσεις. Πρώτα απ' όλα, κάποιες από τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πολύ επικοδομητικές για την υποστήριξη της ανθεκτικότητας, resilience, της αντοχής, ε, προστασία των κέριων υποδομών, προστασία των πολιτικών για την ε, πληροφόρηση, αλλά και διαχείριση κρίσεων. Ουσιαστικά τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια βλέπουμε αρκετές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και που έχουν πάει αρκετά μακριά στην υποστήριξη της αντοχής ή ανθεκτικότητας των επιμέρους κρατών μελών. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο και αφορά το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η κινητήρια μηχανή για πολλές μικρομεσαίες, ε, μικρομεσαίων διαστάσεων, πολλά κράτη-μέλη. Τα περισσότερα κράτη-μέλη βρίσκουν μεγάλες δυσκολίες πολιτικά να αναπτύξουν τέτοιες ε, πρωτοβουλίες αν δεν υπήρχε το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προαγάγουν αυτά τα θέματα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο κενό μεταξύ του δυναμικού των τριών μεγάλων ή των τριών συνενός ε, των μεγαλύτερων αυτών χωρών και των υπόλοιπων ε, μικρότερων χωρών. Έχουμε έναν σημαντικό αριθμό των κρατών μελών που δεν έχουν καν αρχίσει να αντιμετωπίζουν σοβαρά αυτά τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, κάποιες ε, από τις επιδόσεις ε, στο, στην προστασία του κυβερνοχώρου δείχνει το τι γίνεται στην, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δώσω ένα παράδειγμα, η πιο ενδιαφέρουσα ομάδα είναι η European Governance Research Group. Βλέπουμε υψηλού επίπεδου ε, ομάδες που μπορούν να αντιδράσουν άμεσα και που δεν αποτελούν μέρος κάποιου επίσημου, κάποιας επίσημης δομής ή επίσημης οργάνωσης. Και αυτό είναι σημαντικό. Για να είναι κανείς μέρος, μέλος αυτής της οργάνωσης πρέπει να είναι πολύ ικανός στις επιδόσεις του και έχουν λοιπόν κριτήρια ποιοτικά που είναι πάρα πολύ αυστηρά πραγματικά αν υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό κύβερνο ενδεχόμενο, επίθεση ή σύγκρουση, είναι οι καλύτερες ελπίδες μας αυτές οι ομάδες να αντιδράσουμε και δεν θα βοηθούσε να γινόταν ένα ε, θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου όλοι θα είχαν αυτόματα πρόσβαση σε αυτό. Όπως ε, αναφέρθηκε σε σχέση με πέρσι, δεν υπάρχει κέντρο για την κυβερνοπολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει ένα θεσμικό όργανο, ένα γραφείο ή ένα άτομο που να έχει την επισκόψη του τι συμβαίνει από τα τόσα που συμβαίνουν και που είναι πάρα, πολύ, ε, πολλά. Είναι χαμηλό, όχι μόνο χαμηλό, πάρα πολύ χαμηλό το επίπεδο για την ε, κυβερνοασφάλεια από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι τα όσα συμβαίνουν είναι μόνο ε, η κορυφή του παγόβουνου. Τα υπόλοιπα τα οποία δεν είναι γνωστά και δεν διαχέονται και δεν ε, γνωστοποιούνται είναι πολύ περισσότερα και η κίνηση, η δημιουργία task force ε, ή της πρώτης ομάδας, ε, πρώιμης ομάδας μελέτης για αντίδρασης είναι σημαντικά στοιχεία παρότι υπάρχει, ε, υπάρχουν σημαντικοί πόροι που διατίθενται, η δυνατότητα ανταπόκριση ε, δεν είναι ισχυρή, είναι ε, αποδυναμωμένη. Δεν αναφέρομαι μόνο σε σχέση με τον αριθμό των στελεχών που συνεργάζονται, αλλά δεν έχει γίνει κατανοητό το περί τίνος πρόκειται σε σχέση για παράδειγμα με την εξωτερική πολιτική. Α μην ξεχνάμε ότι ό,τι αφορά αυτή την διακυβέρνηση θα έχει επιπτώσει στι επόμενε δεκαετίε. Δεν διαδραματίζει ρόλο η κυβερνοασφάλεια στην ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ε, βλέπουμε ότι γίνεται η προσπάθεια να υπάρξει ανάπτυξη δικτύων ε, ηλεκτρονικών υπολογιστών και δεδομένων, όμως με πολύ βραδείς αργούς ρυθμούς και δεν υπάρχουν άλλα πράγματα που παράλληλα να εξελίσσονται στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ. Και εδώ αυτό είναι σημαντικό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η δράση για τον κυβερνοχώρο. Από την άλλη πλευρά για την Επιτροπή Πολιτικής Ασφάλειας ε, ή για άλλες επιτροπές ε, δεν υπάρχει ε, πρόσβαση στο να ενταχθούν ή να δράσουν στην κυβερνοασφάλεια. Αυτή τη στιγμή η πιεση δεν ασχολείται με την κυβερνοασφάλεια. Είναι, βλέπετε εκτός του πλαισίου της ΚΕΠΑ και για την ΚΟΣΗ το νέο αυτό εσωτερικό σώμα. <clears throat> Δεν είναι απόλυτα σαφές αν αυτό εντάσσεται. Στόχος είναι να εντάσσεται, όμως βλέπουμε ότι θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη αυτό το φάσμα το οποίο απουσιάζει σήμερα και να πρέπει να, να, θα πρέπει να καλυφθεί. Δεν είναι μόνο ε, και θέμα οικονομικό. Οι ελλείψεις αυτές από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προφανής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, λάβει υπόψη και την εμπλοκή των μη κρατικών ε, τομέων. Για παράδειγμα των ομάδων για τις οποίες έκανε λόγο η Χέλη πιο πριν. First, οι άλλες ομάδες που διεθνώς δραστηριοποιούνται και πρέπει να εμπλακούν και να συμμετάσχουν αν θέλει κάποιος να κατανοήσει τι πτυχέ ε, ε, των κυβερνοδραστηριοτήτων και της ε, κυβερνοασφάλειας, εντάσσοντάς σε μια πολιτική ασφάλειας. Κάτι το οποίο χρειάζεται επεξήγηση είναι το hardware attack που αφορά γενικού τύπου επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, που είναι το πιο επικίνδυνο είδος επιθέσεων που γίνονται αναφέρονται σε ατομικά, ε, ατομικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται όπως microchips ή προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις επιθέσεις αυτές και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προστασίας. Είναι σχεδόν αδύνατο να, ε, μπορεί κανείς απόλυτα να ε, προστατεύεται από τέτοιες επιθέσεις. Δεν υπάρχει ε, δυνατότητα να είναι κανείς απόλυτα προστατευμένος. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι, μη κρατικοί τομείς πρέπει να εμπλακούν. Είναι κάτι το οποίο αφορά τις, την προστασία μας. Ωστόσο, είναι ένα θέμα τεράστιας σημασίας και αμφισβητώ αν αυτό έχει γίνει κατανοητό ευρέω ε, στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ένα τεράστια σημασία θέμα. Εφόσον δεν κατανοούμε τα στοιχεία του hardware attack και όλε τι λεπτομέρειε του φάσματο, δεν θα μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Μπορούμε να ε, σκεπτόμαστε την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματο, όμω ε, το hardware των κυβερνοεπιθέσεων είναι ένα πάρα πολύ μεγάλη σημασία θέμα πρέπει επίσης να αποτελέσει αντικείμενο μιας ακρόασης. Ουσιαστικά Έχουμε δύο νομικά μέσα που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν σε περίπτωση ε, κυβερνοεπίθεσης. Το άρθρο 42.7 και το άρθρο 222 όσον αφορά και την αμοιβαία αρρωγή. Και οι δύο αυτές ρήτρες και τα δύο αυτά άρθρα έχουν περιορισμούς που επιβάλλονται. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να βρισκόμαστε επίσημα σε έναν δεδηλωμένο πόλεμο <clears throat> πράγμα το οποίο είναι απίθανο να συμβεί ακόμα και στην περίπτωση σοβαρότατων κυβερνοεπιθέσεων. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να υπάρχει καθορισμένη πράξη τρομοκρατίας. Καθορισμένη πράξη τρομοκρατίας είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Παράδειγμα, οι επιθέσεις στην Εστονία δεν καθορίστηκαν τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τρομοκρατικές πράξεις. Αυτό σημαίνει με άλλα λόγια ότι δεν, έχουμε, δεν έχουμε νομικά μέσα για να υποστηρίξουμε την Εστονία. Μπορούμε να την υποστηρίξουμε μέσω αμοιβαίας προσπάθειας αρρωγής. Δεν έχουμε υψηλού επίπεδου νομικά μέσα ή εργαλεία για να ε, ε, ενθαρρύνουμε να, να παράσχουμε αυτή την αρρωγή. Και αυτό είναι ένα εμπόδιο. Υπάρχουν και άλλα νομικά θέματα εδώ που μπορούμε να επανέλθουμε στι ερωτήσει, ε, όταν θα έχουμε τον χρόνο ερωτήσεων σε αυτά. Επόμενη διαφάνεια. κάποιε από τι συστάσει σε αυτό το πεδίο. Πρώτον και πιο σημαντικά προ όλα τα θεσμικά όργανα. Κατεπηγόντω απαιτείται το επίπεδο πληροφόρηση ε, να είναι δεδομένο ε, ώστε να αυξάνεται η δυνατότητα προστασίας και βλέπουμε ότι τα επίπεδα αυτά είναι πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας τεχνικός όρος αυτός ε, που συμπεριλαμβάνει τα πάντα από την χρήση κωδικών ε, και αλγορίθμων για την προστασία ως την αποθήκευση των δεδομένων και το επίπεδο ε, υλοποίησης αυτών των μέτρων τα ίδια αυτά τα μέτρα είναι σχετικά καλά όμως δεν υλοποιούν, δεν εφαρμόζονται και αυτό συμπεριλαμβάνει και μέχρι πολύ πρόσφατα την, την δυνατότητα να έχουμε μια ομάδα άμεσης ανταπόκρισης μέσω μιας μιας ειδική ομάδας ε, ε, δράσης. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Αυτό λοιπόν στο οποίο προχωρήσαμε είναι ένα πρώτο βήμα και πρέπει να δοθεί συνέχεια. Δεύτερον, αφορά όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στη μελέτη αυτό. Πρέπει ταχαίως να υπάρξει διεύρυνση της διαπίστευσης όσον αφορά θέματα ασφάλειας. Ε, Πολλέ ομάδε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω για παράδειγμα από πλευρά γενική διεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι πολύ ικανές ομάδες, πολύ ικανά στελέχη και έχουν και ομάδες με κάποιους λίγους ανθρώπους ε, που έχουν κάλυψη ε, διαβάθμισης ασφάλειας. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται όμως αυτές οι επιθέσεις, είναι διαβαθμισμένου επίπεδου, ε, δηλαδή ουσιαστικά απόρριτα θέματα και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη διαπίστευση και στην δυνατότητα να ενημερώνονται περισσότερα άτομα ώστε να μπορούν να είναι σε επίπεδο ασφάλειας σε ετοιμότητα. Αυτό αφορά τα θεσμικά όργανα. Επίσης ενθαρρύνουμε, ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη ανταλλαγή αλλαγή πληροφοριών σε ιδιωτικές και κρατικές εταιρικέ σχέσεις σε ευρύ πλαίσιο, ώστε κάθε θεσμικό όργανο να μπορεί να καθορίζει τι σημαίνει για λογαριασμό του αυτό το πράγμα, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ένα παράδειγμα, και πάλι από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρξε η ομάδα EP3R, ομάδα για την ε, αντιμετώπιση και την ανθεκτικότητα ε, του κυβερνοχώρου. Μπορούμε να επεκτείνουμε αυτέ τι δράσει. Υπάρχουν αρκετέ πτυχέ που μπορούν ε, να τύχουν εξέλιξη ε, και να αναπτυχθούν ε, από κοινού ή ξεχωριστά. Πρέπει να θυμόμαστε γενικά στην Ευρώπη ότι τα κράτη-μέλη ξεχωριστά αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα. Κάθε χώρα θα έχει δηλαδή PPP που θα αφορά τον δημοσιονομικό τομέα, τον δημόσιο τομέα, τον ενεργειακό τομέα. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το PPP σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και χρειάζεται, πρέπει να γίνει αυτό. Δεν ενεργούν εν στεγανό ή ε, μέσα σε κάποια κενά ε, οι μονάδε χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει λοιπόν να μπορούν να έχουν αυτές τις πληροφορίες. Πρέπει να τακτοποιήσουμε και να καθορίσουμε τον ρόλο του PSC, COSI και της ε, ομάδας του Συμβουλίου. Δεν υπάρχει σαφής διεργασία ποιος ενημερώνει, ποιοι ενημερώνονται, με ποιο τρόπο εξελίσσεται η πληροφόρηση. Όπως είπα, η ε, ομάδα για την ασφάλεια του Συμβουλίου είναι υπεύθυνη για αυτά τα θέματα και αυτό παραμένει εκτός του πλαισίου της ΚΕΠΑ κι όμως ενθαρρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλες τις ακροάσεις ε, να δρομολογηθούν δράσει ε, για τι σοβαρέ κυβερνοεπιθέσει εις βάρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξαν πολλά επεισόδια τα οποία δεν, ε, για τα οποία δεν, υπήρξαν, δεν υπήρξε ενημέρωση και δεν υπήρξε διάδοση πληροφοριών. Το πρόγραμμα διεύρυνσης για την ενημέρωση των Ευρωβουλευτών είναι σημαντικό. Χρειαζόμαστε όμω μια πολύ ευρύτερη βάση για τη γνώση και διάχυση των γνώσεων, για τις πραγματικές, τα πραγματικά δεδομένα και το ποιοι εμπλέκονται σε όλα αυτά και θα πρέπει να γίνουν ακροάσεις ώστε να αποσαφινιστούν αυτές οι πτυχές. Επίσης ενθαρρύνουμε την χρηματοδότηση των κυβερνομέσων για την κυβερνοασφάλεια και αυτό επειδή είναι δύσκολο να ενταχθούν όλα αυτά σε ένα πλαίσιο. Για παράδειγμα, εμείς ε, από πλευράς μας ε, σε ένα δέκατο της Γερμανίας ως μέγεθος αν έχει για παράδειγμα η Γερμανία 100.000 ε, ε, στρατιώτες και η Αυστρία θα είχε κατά 10.000 αυτό δεν ισχύει κατά αναλογία ε, εκμεταφοράς για την κυβερνοασφάλεια. Χρειαζόμαστε για μικρότερες χώρες πρέπει να δούμε το κόστος για την κυβερνοασφάλεια που είναι πολύ υψηλότερο από ότι στις μεγαλύτερες χώρες και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο οι μικρότερες χώρες ανταποκρίνονται με βραδύτερους ρυθμούς και δεν μπορούν να καλύψουν αυτές όλες τις δαπάνες. Θα πρέπει να εξεταστεί αυτό αυτό, να ότι έχει, μια και έχει συμφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τι χώρε αυτέ, να αναπτύξουν το δυναμικό του για την κυβερνοασφάλεια. Επαναλαμβάνω την έκκληση α, των προελλαλισσάντων. Χρειαζόμαστε ένα συντονιστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα κυβερνοασφάλεια. Κάποιον που θα είναι υπεύθυνο και θα μπορεί να συντονίζει όλε αυτέ τι πρωτοβουλίε και δραστηριότητε και θα είμαστε έτσι πιο αποτελεσματικοί μέσα στο πλαίσιο τη ε, ΚΕΠΑ. Επίση υποστηρίζουμε και ε, επανερχόμαστε σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος Καμιά φορά είναι ασαφές ε, γιατί αυτό δεν έχει παγκόσμια επικυρωθεί. Δεν, είναι, δεν μπορεί να δοθούν απαντήσεις ε, εύκολα. Όμως είναι το καλύτερο μέσο που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή και πρέπει να κυρωθεί για να μπορούμε να δράσουμε πιο αποτελεσματικά. Έχουμε και ένα ρόλο από πλευρά μας ε, μέσα στο πλαίσιο της Επιτροπής για την Ασφάλεια για τον Κυβερνοχώρο. Πρέπει να αναβαθμιστεί όμως αυτό το επίπεδο διότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο, είναι πολύ σύνθετο το επίπεδο των θεμάτων Επίσης υποστηρίζουμε την επικαιροποίηση της ε, αλυσίδας ε, τροφοδότησης ε, όσον αφορά τις επιθέσεις κυβερνοχώρου σε οποίες προαναφερθήκαμε. Η ΕΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία έχουν ε, προγράμματα για την διασφάλιση αυτής της ε, αλυσίδας πληροφόρησης. Στις ΕΠΑ υπάρχουν ε, και συγκεκριμένες εταιρείες που παράγουν μόνο microchips υψηλού επίπεδου, απόλυτα εξειδικευμένα. Στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού υπάρχουν ήδη στόχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κέρια στοιχεία όπως τα microchip δεν θα μπορούν να μολυνθούν με ιούς. Αλλά δεν είναι δυνατόν να είναι κανείς απόλυτα ε, προστατευμένος ε, από τέτοιες επιθέσεις. Επίσης θα θέλαμε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή με μη κράτη-μέλη για το κυβερνοχώρο για να μάθουμε και δάγματα, να αντλήσουμε δάγματα ή να αντλήσουν ε, εταίροι. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας Συνεργασία με τη ΣΥΠΑ που είναι πάρα πολύ καλό και πρέπει να βρούμε, υπάρχουν και άλλε χώρε με τι οποίε έχουμε μηχανισμού συνεργασία. ή πρέπει να βρούμε, πρέπει να δούμε παραδείγματο χάρη τι μπορούμε να κάνουμε με τη Ρωσία, την Κίνα, την ε, Ινδία. Θα έπρεπε όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό να έχουμε στενότερους ε, δεσμού. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν κάποια μέσα χρηματοδότησης για τη στήριξη της κυβερνοασφάλειας. Σε κάποιες χώρες όπως τη Γερμανία υπάρχει ένα ειδικό γραφείο για την κυβερνοπροστασία και υπάρχουν δωρεάν εργαλεία πάρα πολύ αποτελεσματικά τα οποία προωθούνται για την διαχείριση κινδύνων, για τη βασική προστασία ε, και είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, καλύπτουν ένα πολύ μικρό τμήμα βέβαια του πιθανού ε, της πιθανής εμβέλειας εργαλείων πληροφορικής ή διαχείρισης κινδύνων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει κάποια προγράμματα. Δεν θα αναφέρω μάρκες, ε, εμπορικά σήματα, αλλά υπάρχουν προγράμματα λογισμικού που είναι ελεύθερα ε, για χρήση οικιακή μέχρι στιγμή. Θα μπορούσε κανεί να τα μεταφορτώσει, να, χρήσει, να τα χρησιμοποιεί ε, στο σπίτι του, αλλά οι εταιρείε πρέπει να τα πληρώσουν για να τα αποκτήσουν τι κάνουν τώρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, μπορούν να τα κατεβάσουν και να τα χρησιμοποιήσουν αυτά τα προγράμματα δωρεάν. Ίσως θα έπρεπε να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία προγραμμάτων ε, που θα έχουν μια άδεια γενική και θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό για να προστατευτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από κυβερνοεπιθέσεις. Επίσης, σίγουρα επιγόντως πρέπει να μιλήσουμε για ένα κυβερνοθεματολόγιο ε, στην ΚΕΠΑ, στην Επιτροπή, στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Επίσης, να πούμε τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτό το κυβερνοθεματολόγιο. Ε, πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τη διαδικτυακή διακυβέρνηση που είπαμε ότι πρώτα απ' όλα σημαίνει πώς ορίζουμε σε πολιτικό επίπεδο την πραγματικότητα επίση κωδικού του διαδικτύου. Δεν μπορεί κανείς σε καμία περίπτωση να ε, έχει ε, επιτυχία και να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα εάν δεν το κάνει αυτό. Ό,τι αποφασίσουμε τώρα θα καθορίσει την πορεία μας ε, και την πορεία του διαδικτύου για τα επόμενα 5-10 χρόνια αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας ίσως ή οποιασδήποτε μελλοντικέ ενδεχόμενες κυβερνοσυγκρούσεις. Όλα αυτά βασίζονται στις αποφάσεις που θα ε, ληφθούν από σήμερα αλλά δεν βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά. Το ίδιο ισχύει με τη συμμετοχή σε διεθνείς συζητήσεις για την ανάπτυξη των προτύπων για τις κυβερνοσυγκρούσεις. Έχουν γίνει συζητήσεις κυρίως σε επίπεδο ΟΗΕ και ΟΑΣΕ όπως είπε η συναδελφός μου πριν. Όλες αυτές οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη κοινών συμφωνιών μεταξύ των χωρών χωρών για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται στον κυβερνοχώρο. Βέβαια δεν θα έχουμε μια σύμβαση της Γενέβη για τον κυβερνοχώρο σύντομα, ούτε μια συνθήκη ελέγχου των ε, εξοπλισμών, γιατί δεν μπορεί κανεί ούτε να την ε, επιβάλλει να την ελέγχει. Αλλά θα μπορούσαμε όμω να συμφωνήσουμε για τα πρότυπα, τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν, είτε θα πρέπει, ή τι θα πρέπει να κάνουν οι χώρε. Αυτέ οι συζητήσει ε, συνεχίζονται για τουλάχιστον ένα χρόνο, ενάμιση περίπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ δεν διαδραματίζει και κανένα σπουδαίο ρόλο οι σημαντικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν δεν ε, προάγονται. Αλλά περί αυτού πρόκειται. Αυτές οι σημαντικές αρχές είναι. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης είναι ένας τομέας που απασχολεί ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ο κυβερνοχώρος ε, ε, τρεις ε, μήνες ε, ισχύει σχετική υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πάρα πολύ μικρός χρόνος στον κυβερνοχώρο. Πάντως πρέπει να ενθαρρυνθεί η πρωτοβουλία αυτή όσο η στρατιωτική συνεργασία, η αστυνομική συνεργασία, τόσο σημαντική πρέπει να θεωρείται και η κυβερνοασφάλεια. Θα πρέπει λοιπόν και η υπηρεσία εξωτερική δράση να μπορεί και στι αποστολέ τη αλλά και στι Βρυξέλλε να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Επίση, θα πρέπει γενικά να αξιολογήσουμε την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις. Πρέπει να υπάρχουν παράμετροι ε, πώς θα μπορεί κανείς να αντιδράσει σε μια κυβερνοεπίθεση, αλλά να υπάρξει και μια δεξαμενή προβληματισμού γενικότερα, μια ομάδα προβληματισμού. Ε, αν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει σοβαρή κυβερνοεπίθεση σε μία περισσότερες χώρες ή σε έναν περισσότερους οργανισμούς και αν μπορεί πολιτικά να κάνει κάποιες δηλώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως αρκεί ως πρώτο βήμα. Πρώτα απ' όλα βέβαια θα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνο, να δούμε ποιος αναλάβει την πολιτική ηγεσία. Επίσης πρέπει να υπάρξει καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων πρωτοβουλειών της Κομισιόν σε επίπεδο ΚΕΠΑ και ξανά στην ΚΕΠΑ γιατί υπάρχουν πολλοί αρμόδιοι, είναι μεταξύ αυτών και η γραμματεία του Συμβουλίου. Υπάρχουν ε, ε, δυσκολίες στο συντονισμό. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ασχολούνται με, την ΚΕΠΑ αλλά δεν γνωρίζουν όλα όσα γίνονται και καλό θα, έπρεπε, καλό θα ήταν υπάρχει μια γενικότερη επισκόπηση. Επίσης με την EUMC θα πρέπει να υπάρξει στήριξη για τη σύσταση κοινών ε, πλαισίων πολιτικής έχουν ξεκινήσει σχετικές προσπάθειες, πρέπει να συνεχιστούν. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι πόροι ιδίω ε, στο πλαίσιο της Γραμματείας του Συμβουλίου και της ΕΙΕΔ, αλλά και στην ίδια την Κομισιόν. Λίγοι, πολύ λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Ε, επί του παρόντος, κατά την άποψή μου περισσότεροι είναι στην υποομάδα της ΓΔ αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν κατανόηση για αυτά τα θέματα παρότι εργάζονται εδώ και καιρό με αυτά. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να διευρύνουμε τον αριθμό των ατόμων οι οποίοι από αναλυτική πλευρά μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα και να βελτιώσουμε επίση και τι δυνατότητε που έχουν να επικοινωνούν μεταξύ του. Αυτή είναι η βασική στόχη ε, και το σύστημά του, αν δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνία, είναι αυτό το οποίο θα δεχθεί πρώτο την επίθεση. Άρα, αν δεν υπάρχει επικοινωνία και αντιμετώπιση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επίση, ε, νέε πρωτοβουλίε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα. Υπάρχουν διαφορετικέ πρωτοβουλίε, τι οποίε διερευνούν ε, οι ερευνητικοί οργανισμοί στον τομέα της άμυνας στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη ΣΥΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και βέβαια εδώ έχουμε το πρόβλημα ότι τα μικρά ή μικρομεσαία κράτη δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία, σε αυτήν την έρευνα. Και αυτό το χάσμα θα διευρύνεται όλο και περισσότερο αν δεν γίνει κάτι. Επίση, θα πρέπει να δούμε και τι διεθνεί οργανώσει, του διεθνεί οργανισμού που δραστηριοποιούνται επί του παρόντο στον τομέα αυτό. Από πλευρά ΚΕΠΑ, για παράδειγμα. Να δούμε τι μπορεί να κάνει Έχουμε πολλά πράγματα τα οποία ε, διακυβεύονται και διμερός και πολυμερός. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, γιατί αν δεν ξέρουμε ποιε είναι οι προκλήσει, δεν θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό λοιπόν είναι και ε, ουσιαστικά το τέλο τη παρουσίασή μα. Ε, είμαστε βέβαια στη διάθεσή σα και για ερωτήσει. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε λοιπόν τώρα έναν γύρο έρωτα απαντήσεων και μετά θα έχουμε και το δεύτερο πάνελ. Παρακαλώ, ο κύριος Γκάλερ. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διερωτώ με ότι ε, για όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι καινούργια για μένα θα έλεγα και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η, η, η ομιλία αυτή που ακούσαμε, αλλά ήθελα να ξέρω πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι, δηλαδή μια επίθεση τι, που θα οδηγούσε, ε, θα είχαμε... Πώς ορίζεται η σοβαρότητα. Υπάρχουν και κάποια κριτήρια τα οποία αποφασίστηκαν από ό,τι ξέρω. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω εσείς ε, τι πιστεύετε, πότε μια επίθεση στον κυβερνοχώρο μπορεί να θεωρηθεί ως μια πολεμική ε, ενέργεια και ε, θα πρέπει να, ας πούμε, να γίνει μια επίθεση με στρατό σε μια χώρα, να, πότε θα υπάρξει διέλευση συνόρων τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά επίσης και για τις δύο εισηγήσεις από τους δύο προσκεκλημένους. Είδαμε από αυτές τις εισηγήσεις ότι βρισκόμαστε εδώ σε ένα πολύ περίπλοκο σύνθετο περιβάλλον. Ξεκίνησε ήδη με την πρώτη διαφάνεια, με την πρώτη διαφάνεια όπου το είδαμε ότι δεν υπάρχει ούτε καν κοινό τρόπος ε, καταγραφής ε, με τους τίτλους και τα ονόματα και αυτό είναι χαρακτηριστικό όταν κάνουμε λόγο για το, το κυβερνοέγκλημα, κυβερνοασφάλεια, κυβερνοπόλεμο ή οτιδήποτε συναφές και αυτό συσχετίζεται επίσης με το ότι μέσω του διαδικτύου όλες οι σφαίρες παν, παγκοσμίως, η ιδιωτική σφαίρα της ιδιωτικής ζωής αλλά και κάθε άλλη σφαίρα, κάθε θέμα μπορεί να αποτελεί αντικείμενο πρόσβασης. Κάθε ένας μπορεί να είναι θύμα ή αντικείμενο επίθεσης. Και αυτό αφορά και την εξωτερική ασφάλεια, εσωτερική ασφάλεια, την άλλη πλευρά, πρόκειται για οικονομικό έγκλημα, οικονομική εγκληματικότητα ή ιδιωτική αντιπαράθεση και τριβές μεταξύ ιδιωτών ως ατόμων. Και εξου και αυτή η εισήγηση και τα θέματα τα οποία τίθενται για πολλούς από εμάς σε πολλά επίπεδα στο Ευρωκοινοβούλιο είναι πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και εμείς εδώ στην δική μας επιτροπή, στη δική μας υποεπιτροπή για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, καλούμεθα να δράσουμε. Και φυσικά σε αυτά τα θέματα που αφορούν αυτές τις σφαίρες που περιέγραψα για την κοινή ασφάλεια, την εξωτερική ασφάλεια, εσωτερική ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι τα πιο σημαντικά. Και εξού και οι ερωτήσεις που διατυπώνω και πρέπει να διατυπώσω και που αναφύονται και που δεν υπάρχουν φυσικά ακόμα κάποιες απαντήσεις έτοιμες, κομμένες και ραμμένες. Είπατε ότι μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες είναι να διαπιστωθεί από ποιον προέρχεται μια τέτοια επίθεση. Ποιος είναι ο υπεύθυνο για μια τέτοια επίθεση. Είναι μεγάλη διαφορά αν είναι κάποιο hacker ω ιδιώτη, ω άτομο, ή αν είναι κάποιο που από μια κυβέρνηση, από ένα κράτο έχει εντολή να, κάνει, να διαπράξει αυτέ τι επιθετικέ ε, πράξει που παρισφρέουν και πλήττουν το σύστημα μιας άλλης χώρας και το παραλύουν ενδεχόμενα. Είτε πρόκειται για δίκτυο ε, ηλεκτρικής ενέργειας, ε, ηλεκτρικού ρεύματος ή στρατιωτική σταθμή ή πλήγματα στο στρατιωτικό τομέα. Άσχετα, ξεκινούν πάντα με αυτά τα προβλήματα τα οποία προανέφερα. Και η ερώτηση που διατυπώνω ίσως θα ήταν ένας τρόπος να βρίσκαμε τρόπους αντίδρασης νόμιμα και θεμητά να αντιδράσουμε και να ανταποκριθούμε. Θα ήταν ένας τρόπος να καθορίσουμε Ποιο είναι εκείνος εναντίον του οποίου στρέφεται μια τέτοια επίθεση. Αν πρόκειται για μια επίθεση εναντίον στρατιωτικών στόχων ή όσον αφορά την ασφάλεια, θα πρέπει με τους ίδιους, με τα ίδια μέσα να είναι θεμητό να αντιδράσει κανείς, να οδηγηθεί σε πλήγματα που θα δώσει στον επιτιθέμενο και με αυτά τα μέσα όταν έχουμε σε παράλληλο τομέα οικονομικό έγκλημα ή παράλληλες οικονομικές ε, ε, πρωτοβουλ... Ε, πλήγματα εις βάρος οικονομικών συμφερόντων πάλι θα έπρεπε να υπάρχει νομιμοποίηση να αντιδράσει κανείς και να πλήξει τον εχθρό του με αυτόν τον τρόπο ή να προσφύγει σε ένα δικαστήριο λόγω ζημιάς που έχει υποστεί. Όλο αυτό το φάσμα το αναφέρω ως δυνατότητα. Αυτό θα ήταν μια δυνατότητα δυνατότητα προσέγγισης, δυνατότητας ε, θεμητής ε, ανταπόδοσης. Και ένα άλλο ερώτημα, όταν έχουμε το τομέα της εξωτερικής ασφάλειας και κινούμαστε σε αυτά τα θέματα, τότε θεμητά ερωτήματα αναφύονται, όχι μόνο για την άμυνα, αλλά και για την ίδια την επίθεση προληπτικές επιθέσεις ας το πούμε έτσι ώστε να μην υπάρξει το χειρότερο παράδειγμα, για ένα πυρηνικό αντιδραστήρα στο Μπουσέρ του Ιράν, για παράδειγμα, όπου εναλλακτική λύση θα ήταν οι συμβατική βομβαρδισμοί ή η πιο λεπτή διαφοροποίηση ε, για τέτοιου είδους ε, πλήγματα να οδηγήσουμε κάτι σε αυτή τη μονάδα, σε αυτόν τον πυρηνικό αντιδραστήρα του Ιράν, ώστε να τον καταστήσουμε αυλαβή, να τον βλάψουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του. Σε αυτό το τομέα, σε αυτό το επίπεδο, τίθεται ερώτημα. Ποιο θα ήταν το νόμιμο ή θεμητό μέσο ανταπόδοσης ή απάντησης για μια τέτοια αναμενόμενη επίθεση, ώστε να μην υπάρξει αυτή η επίθεση, να αποφύγουμε τέτοιο ενδεχόμενο επίθεσης. Αυτό αφορά και την έναρξη της συνεδρίασης όπου στην αρχή ε, ο πρόεδρος της Επιτροπής μας είπε για το θέμα του άρθρου 5 ότι στο ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, ως σημαντική ρήτρα αρρωγής ε, αντιμετωπίζεται και υπάρχουν διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις. Δεν είναι όλοι σύμφωνοι αν μια κυβερνοεπίθεση θα πρέπει να οδηγεί στην δρομολόγηση και δραστηριοποίηση της ρήτρα του άρθρου 5, του εδαφίου του άρθρου 5. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Κοπά, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικαιρή συζήτηση και γιατί συμπίπτει με την ανάληψη σοβαρών πρωτοπλών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για μια νέα πολιτική τη συμμαχία στον τομέα της κυβερνοασφάλεια, αλλά και επειδή όπω είπατε το γεγονός αυτό από μόνο του πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε τι κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο γενικότερο πλαίσιο η παρουσίαση μια ενημερωμένη εκδοχή ε, των ε, εκθέσεων ε, ένισα ε, είναι κάτι το οποίο επίσης ήταν, ε, έγινε σε επίκαιρη χρονική στιγμή. Καλό είναι να αντλήσουμε κάποια κοινά συμπεράσματα από τις εκθέσεις αυτές. Πρέπει να δούμε πόσο προετοιμασμένες είναι οι χώρες για να αντιμετωπίσουν κυβερνοεπιθέσεις. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο αντιμετώπισης αντιμετώπισης των ε, επιθέσεων. Ε, αν δει κανείς τα συμπεράσματα των ε, δύο εκθέσεων που προανέφερα, βλέπει κανείς ότι δεν έχει διαπιστωθεί μεγάλη πρόοδος μετά το 2006 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι μεν αντιλαμβάνεται πως έχει κατάσταση, έκανε και κάποιες προτάσεις από το 2011 και ζητά ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα ε, δίκτυο διαφόρων ομάδων από το 2012 και ζητά περισσότερη συνεργασία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνέ επίπεδο. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πράγματα τα οποία πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν αρκούν όμως αυτά και πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Αυτό το οποίο χρειάζεται κατά την άποψή μου είναι μια πιο συνεκτική, πληρέστερη προσέγγιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει επίσης να αναπτύξουμε δυνατότητες ε, στο επίπεδο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ε, και ε, θα πρέπει κάθε κυβερνοεπίθεση να την αντιλαμβανόμαστε Sorry. Uh, Ω ένα μεμονωμένο συμβάν και θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην πρόληψη και όχι στην αντίδραση σε μια στρατιωτική απειλή. Γι' αυτό μιλάω για δυνατότητε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, δεν θα πρέπει να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη και θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό για αποφυγή επιπλέον κόστου, όπου αυτό βέβαια είναι δυνατό. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Θα μπορούσατε να μα κάνετε μια αντικειμενική εκτίμηση των μέτρων τα οποία ε, προτείνει η Κομισιόν. Τι νομίζετε Τι πιστεύετε για την τρέχουσα κατάσταση. Και επειδή αναφέρθηκα στην Ενίζα αρχίζοντας, ε, θέλω να πω ότι ε, υπάρχει η όλη συζήτηση για το κατά πόσον αυτή η υπηρεσία είναι χρήσιμη και επίσης κατά πόσον θα πρέπει να ξεχρονιστεί ε, Ξέρουμε ότι η εντολή του ΕΝΙΣΑ τον ε, Μάρτιο του 2012 νέη. Εμείς πιστεύουμε στην Επιτροπή μας ότι πρέπει να αναπτύξουμε δυνατότητες κυβερνοπροστασίας. Ε, επομένως πρέπει νομίζω να καταλήξουμε στο ότι είναι χρήσιμος ο οργανισμός ΕΝΙΖΑ γιατί παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και στην Ένωση και στα κρατημέλη και συμβάλλει ε, στην έρευνα για την κυβέρνηση Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Μπουτικόφερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για αυτές τις παρουσιάσεις, τις εισηγήσεις. Ήταν πραγματικά διαφωτιστικές. Έχω πολύ, πολλές περισσότερες ερωτήσεις από αυτές που μπορώ να διατυπώσω. Όμως όλες οι ερωτήσεις ε, κινούνται γύρω από το θέμα της διακυβέρνησης, governance, μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω αφορά τη σχέση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της Ένωσης. Εσείς, αν τα θυμάμαι και τα κατανόησα σωστά, υπό την προοπτική των μεσαίων και μικρότερων χωρών αναφέρατε κάτι και είπατε ότι πρέπει ιδιαίτερα να υπάρξει μια απάντηση κοινή για αυτές τις χώρες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η δεδομένη προθυμία και βούληση των μεγαλύτερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεισφέρουν ενεργά ώστε να δημιουργηθεί μια τέτοια κοινή ας το πω έτσι, προσέγγιση και να ενταχθούν και να ε, ολοκληρωθούν οι προσπάθειες των μικρότερων χωρών ή μεσαίων χωρών σε αυτό το πλαίσιο. Δεύτερον, στις δικές σας παρουσιάσεις, με τα δικά σας λόγια, παρουσιάστηκε το πρόβλημα του πόσο θα μπορούσε να είναι επιτυχές τα θέματα της κυβερνοασφάλειας αποκλειστικά ή κυρίως υπό στρατιωτικό πρίσμα να εξετάζονται και να διαχειρίζονται. Από αυτό απορρέουν και θέματα διακυβέρνησης ή διαχείρισης. Κατά πόσον μπορεί θεμητά να οδηγηθούν όλα αυτά σε ένα Υπουργείο Άμυνα ή σε ένα Υπουργείο Εσωτερικών ή στον Υπουργό Εσωτερικών ή Υπουργό Άμυνα. Κατά πόσον υπάρχουν τέτοια χειροπιαστά α το πω, στοιχεία που να οδηγούν σε μια τέτοια πορεία. Και αντίστροφα, στο ρωσικό και στο κινέζικο υπόδειγμα ή παράδειγμα αναφέρθηκε ο ρόλο των hacker communities, των ομάδων επιδρομέων του κυβερνοχώρου. Υπάρχουν κάποια στοιχεία από την πείρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αναφέρθηκε τίποτα αν θυμάμαι εγώ καλά. Πώς δηλαδή η κοινότητα των hackers στην Ευρώπη μπορούν να εντάσσονται μέσα σε αυτό το θέμα ή πώς θα μπορούσαν αυτοί οι hacker να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο ή όχι. Το ΝΑΤΟ και η ΚΕΠΑ είναι εδώ ένα ερώτημα το οποίο αναφύεται. Ποιες προσεγγίσεις υπάρχουν για συνεργασία ή και διπλοεπικαλύψεις μεταξύ αυτών των δύο θεσμικών οργάνων ώστε να αποφύγουμε να μην υπάρχουν τέτοιες διπλοεπικαλύψεις έργου μεταξύ τους και επιπλέον όταν περιγράφηκε η κατάσταση της, της Κίνας και της Ρωσίας όταν αναφέρθηκε η Κίνα και η Ρωσία κατά κάποιο τρόπο με σαφήνεια χαρακτηρίστηκαν ως χώρες adversarial nature, δηλαδή θα έλεγα όχι εχθροί αλλά αντίπαλοι εντό εισαγωγικών. Αυτό ίσω συμπίπτει και με τα βιώματά μας και τα στοιχεία που έχουμε. Όμως με ποιο τρόπο, με ποιο τρόπο ίσως υπάρχουν από τη δική σα πείρα κάποια στοιχεία που να δικαιολογούν στρατηγικέ communality κοινών χαρακτηριστικών ή στοιχείων. Γιατί και αυτές οι χώρες ε, μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επιθέσεων κάποιων hacker Κατά πόσον λοιπόν υπάρχει έστω η προσέγγιση μιας βάσης συνεργασίας με βάση διεθνείς προδιαγραφές με τον περίγυρο αυτών, με αυτές τις χώρες. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό, τελευταία ερώτηση. Αναφέρατε resilience, ανθεκτικότητα ή αντοχή και deterrence, αποτροπή, ως ιδανικά για την, ως, ως στοιχεία αντίδρασης. Και περιγράφηκε η περίπτωση των ΙΠΑ που βασίζονται στο χαρτί του της hard deterrence, της σκληρής ομής αποτροπής. Χρησιμοποιήθηκε αυτό το χαρτί από τη ΣΥΠΑ και λειτουργήσε αυτή η μέθοδος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Herrenhauser, σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ θερμά για αυτή την περιεκτική μελέτη. Πολύ καλές προσεγγίσεις για αυτό το θέμα δίνονται. Ένα πράγμα το οποίο είδα να απουσιάζει και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού είναι το θέμα των δαπανών. Η αναφορά σε δαπάνες και κόστη. Θα με ενδιαφέρε, υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, υπάρχουν κάποιοι πίνακες. Τι συνεπάγεται το κυβερνοέγκλημα και οι κυβερνοεπιθέσεις ως δαπάνες, ως επιπτώσεις, συνέπειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη πλευρά τι επενδύουν χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία ή σε σχέση με τη ΣΥΠΑ για την κυβερνοασφάλεια. Ίσως υπάρχουν κάποια ποσά, κάποια στοιχεία ώστε να εντάξουμε καλύτερα αυτό το πλαίσιο στις συζητήσεις μας. Επόμενο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας, τις τόσο λεπτομερείς. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω που συνδέονται με το σύστημα πρόληψης. Στον τομέα αυτό, έστω και αν δεν έχουμε έναν συμφωνημένο ορισμό του κυβερνού εγκλήματος, που είναι μια ενέργεια, μια διαδικασία κτλ. κτλ πιστεύω ότι η προσέγγιση της πρόληψης είναι πιο κατάλληλη. Μπορεί, μήπως εσείς έχετε να μας προτείνετε κάποιες διαδικασίες που θα οδηγούσαν σε αυτή την πρόληψη και που προέρχονται από την, όχι από τον στρατιωτικό τομέα μόνο, αλλά και από τον επιχειρηματικό κτλ. Και δεύτερο, τι γίνεται με την ποινική δίωξη κατά των υπευθύνων, διότι δεν έχουμε και εδώ μια κοινή προσέγγιση. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν την ικανότητα να διεξάγουν μια ακριβή και λεπτομερή έρευνα για αυτού του είδους τα εγκλήματα διότι δεν υπάρχουν εμπειρογνώμονες, ε, διότι ενδεχόμενο το κράτος να είναι ανίκανο να αφιερώσει ανθρώπινους πόρους στον τομέα αυτό. Το 2008 αποφάσισε το, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο να δημιουργήσει αυτό το, αυτή την πλατφόρμα δεν ξέρω εάν ήδη αυτή η πλατφόρμα πρόληψης ε, έχει δημιουργηθεί στα κράτη-μέλη, γιατί μιλάμε για περισσότερο ε, εγκλήματα κατασκοπίας, αν θέλετε, και εξαρτώνται από την αντίδραση ε, ταχύτητα αντίδρασης των κρατών μελών. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριος Παλέσκη. Ευχαριστώ. Παρακολούθησα την, ε, το περισσότερο μέρος της ομιλίας, αλλά έπρεπε να φύγω γιατί έπρεπε να ψηφίσω σε μια άλλη επιτροπή. Πιστεύω ότι τα κυβέρνο όπλα, αν θέλετε, είναι τα πιο προηγμένα όπλα και η άμυνα στο κυβερνοχώρο είναι η πιο σύγχρονη, αν θέλετε, άμυνα. Και χρησιμοποιούμε όπλα εδώ όπως τα κανόνια και ε, οι θώρακες. Ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τέτοιο παραλληλισμό. Δηλαδή ότι αν κάποιος χρησιμοποιεί μια, μια σφαίρα θα πρέπει και εμείς να βρούμε ένα, μια πανοπλία τέλος πάντων η οποία να μπορεί να αντισταθεί στην, ε, στα όπλα αυτά. Και ρωτώ, η πανοπλία την οποία έχουμε είναι κατάλληλη για την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Μπορεί μια άμυνα στον κυβερνοχώρο να είναι ανίκητη και τώρα σε τι στάδιο βρισκόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σύστημα άμυνας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μάθαμε πάρα πολλές πληροφορίες και εκτιμώ ιδιαίτερα τις ε, παρουσιάσεις που έγιναν. Κάποιες, κάποιοι συνάδελφοι έθεσαν τις ερωτήσεις ε, που ήθελα να κάνω κι εγώ. Εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για τις ε, επιθέσεις, ε, για τις hardware attacks. Αναφερθήκατε στον τεράστιο και άμεσο κίνδυνο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί και διερωτώ με πού, είναι, πού γίνεται η επίθεση στον, στους υπολογιστές, στο hardware, στο software, πού ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις, ε, πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα απαντήσω με τη σειρά και μετά θα δώσω και το λόγο στην συνάδελφο για να ολοκληρώσει τις απαντήσεις όπως εκείνη θεωρεί σκόπιμο. Καταρχάς, όσον αφορά τον κίνδυνο μιας κυβερνοεπίθεσης, πόσο σοβαρή μπορεί να είναι και μετά ποιος είναι ο ορισμός του κυβερνοπολέμου το πόσο κακή, πόσο επικίνδυνη μπορεί να αυτή η επίθεση είναι ένα βασικό ερώτημα το οποίο μας απασχόλησε τα τελευταία 10-12 χρόνια. Από τα άτομα τα οποία ασχολούνται με το θέμα αυτό, να σας πω ότι η επίθεση μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ κακή. Το πρόβλημα είναι μήπως προκαλούμε περισσότερο κακό συζητώντας για το θέμα αυτό και αντί να, αντί να κάνουμε κάτι, να αντιμετωπίσουμε ή μπορούμε να το συζητάμε και βοηθάει η συζήτηση. Ε, υπάρχει ένας κυβερνο, κυβερνοσυζήτηση, αν θέλει, ένας κυβερνοπόλεμος με λόγια αυτή τη στιγμή, όπως λέει και ο Λευκός Και το πρόβλημα είναι να δούμε ποιες είναι, ποια είναι τα πολιτικά κίνητρα ε, για να γίνεται αυτή η συζήτηση γιατί πολλέ φορέ στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ο πόλεμο αυτό των, των λόγων γίνεται ανάμεσα ε, στο Υπουργείο Άμυνα, στι υπηρεσίε κατασκοπία κτλ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, όμω οι επιθέσει στον κυβερνοχώρο μπορούν να είναι πολύ επικίνδυνες, μπορούν να δημιουργήσουν τεράστιες φασαρίες, όπως υπάρχουν διάφορα εφιαλτικά σενάρια, αλλά είναι εφιάλτες. Δεν είναι σαν μια πυρηνική επίθεση βέβαια προφανώς. Υπάρχει όμως ένας παραλληλισμός στον κυβερνοχώρο. Ε, μπορεί να γίνει μια επίθεση στον κυβερνοχώρο όπως μπορεί να γίνει και μια πυρηνική επίθεση. Αλλά ελπίζουμε ότι και τα δύο είναι ε, σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα έχουμε δει πολλέ φορέ στον κινηματογράφο. Όντω μπορούν να συμβούν. Ελπίζουμε ότι δεν πρόκειται να συμβούν. Τώρα, υπάρχουν ορισμοί όσον αφορά την, ε, την, ε, τις επιθέσεις, τις πολεμικές επιθέσεις ε, στο κυβερνοχώρο και πόσο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι γίνεται, υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα σε μια στρατιωτική επίθεση και στον, σε μια επίθεση στον κυβερνοχώρο. Υπάρχει βέβαια και η κατασκοπία στον κυβερνοχώρο ε, μπορεί πολλές φορές ε, πληροφορίες να καταστραφούν, συστήματα να καταστραφούν. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί τελικά πολεμική ενέργεια, πολεμική επίθεση. Τώρα, άλλη ερώτηση για το πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε, πώς μπορούμε να απαντήσουμε και να εντεπιτεθούμε με τα ίδια μέσα. Και η δεύτερη ερώτηση αφορούσε την προληπτική επίθεση. Εγώ μίλησα πάρα πολύ για τα θέματα αυτά, για το πώς μπορούμε να αντεπιτεθούμε αν θέλετε. Και έδωσε και μια συνέντευξη η οποία ε, αναμεταδόθηκε αρκετά. Ας πούμε το IMF ε, υπέστη μία επίθεση από κάποιους που δεν γνωρίζουμε και επομένως γιατί να μην υπάρχει μια σφαιρική, μια οικουμενική απάντηση σε ένα πρόβλημα σφαιρικό και οικουμενικό. Στο, στην περίπτωση του Δουνουτού, του IMF, μπορεί να γίνει μια έρευνα από μη κρατικό φορέα. Ένα συνάδελφο με τον οποίο συνεργαζόμαστε από το θέμα είπε ότι γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε ένα κλέφτη για να πιάσει τον κλέφτη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι Ευρωπαίοι hacker έχουν επιτίθενται στους Ρώσους ή στους Κινέζους ομολόγους τους, αλλά η ικανότητά μας στην, ε, κοινωνία των πολιτών θα ε, μπορεί να, να συνεισφέρει στην, ε, στην άμυνά μας. Δηλαδή να κάνουν κάποιες μελέτες, κάποιες αναφορές όλα τα στοιχεία ε, που αφορούσαν την επίθεση στη Γεωργία και στην Εσθονία ε, προέρχονται από τέσσερις αναφορές, μία από αυτές την έγραψα εγώ, ε, και που προέρχονται από τους πολίτες. Βέβαια υπάρχουν και άλλες πληροφορίες από, τις, ε, από την κατασκοπία κτλ. Όμως ε, οι, εφημερίδες δημοσιεύουν στοιχεία τα οποία προέρχονται από, την, από τους πολίτες ε, που μας ζητούν δηλαδή να πούμε την άποψή μας εάν την άποψη αυτή τη θεωρούν σοβαρή την δημοσιεύουν. Τώρα, οι προληπτικές επιθέσεις. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι υπέρ αυτή τη αντιμετώπιση. Υπάρχει βέβαια και ένα επιχείρημα ότι αν ξέρω εγώ ε, θέλει να βομβαρδίσουμε κάτι θα κάνουμε την επίθεση μέσω κυβερνοχώρου. Εγώ δεν απαντάω σε αυτό το θέμα. Ε, θεωρώ όμως ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Όταν στείλετε ένα πύραυλο κρούζ, ας πούμε, ε, καταστρέφεται και ο στόχος και ε, ο πύραυλος. Εάν βάλεις όμως ε, έναν ιό σε ένα σύστημα, αυτός ο ιός μπορεί να επιστρέψει σε σένα όμως. Και αυτή ήταν μια, ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τις Ηνωμένε Πολιτείες δεν έχουν ε, αρνηθεί ότι έχουν στείλει ιούς ούτως ή άλλως και δεν ξέρω τι να σας πω, δεν, δεν, θέλω να πω την άποψή μου, δεν μπορώ να ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα αλλά ξέρω ότι όσοι ε, έχουν ξεκινήσει τέτοιου είδους ε, ιούς έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα το οποίο θα μας ακολουθεί εδώ και χρόνια. Τώρα, θα έχουμε περισσότερες επιθέσεις σε διεθνέ επίπεδο από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. όντω αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα μπορούσαμε να εξετάσουμε. Τώρα, όσον αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική, ε, δεν, έχουν, δεν έχει γίνει μεγάλη πρόοδο. Αυτό το λέμε ούτω ή άλλω και στι αναφορέ μας. Για να γίνει μια αντικειμενική ε, αξιολόγηση των προτάσεων της Κομισιόν, θα ήθελα να σας ζητήσω να διαβάσετε την έκθεση γιατί εκεί μπαίνουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Όντως ε, πρέπει να γίνει μια απάντηση σε επίπεδο κρατών μελών, δηλαδή θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τις συστάσεις σε τεχνικό επίπεδο όμως πρέπει να δούμε ε, αν έχουν τα μέσα για να υλοποιήσουν τις συστάσεις αυτές, αλλά και από οικονομικής πλευράς θα πρέπει να δούμε έχουν τους πόρους ε, και για την τεχνολογία, αλλά και για τους, ε, τους, και τους ανθρώπινους πόρους να τα κάνουν, να, να υλοποιήσουν τις συστάσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Τώρα για την εντολή για την Ενίζα, όντως είναι, θα πρέπει να καθοριστεί ο ρόλος της στο μέλλον και είναι καθοριστικός ο ρόλος αυτός, θα έλεγα. Η Task Force ε, έχει την βάση της στην, ε, στις Βρυξέλλες, πρέπει να είναι κοντά ούτως ή άλλως Εγώ θα προτιμούσα να είναι στην Αθήνα σε κάποιο νησί η έδρα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι δική μου επιλογή. Ε, πάντως ο ρόλος της ΕΝΙΖΑ είναι να ε, αξιολογεί από μια τρίτη ματιά τις επιθέσεις στην Ευρώπη και ο ρόλος ε, θα, ρόλος θα αυξηθεί στο μέλλον θα έχει να παίξει έναν επιχειρησιακό ρόλο, ρόλο όσον αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών ε, αυτό είναι μια επανάσταση πραγματικά πιστεύουμε, μια καινοτομία, διότι η ΕΝΙΖΑ θα έχει αρμοδιότητες ε, ε, περισσότερες από αυτές που έχουν οι κυβερνήσεις. Γιατί πολλοί λένε ότι όντως η ΕΝΙΖΑ έχει περισσότερες αρμοδιότητες και γνώσεις από ότι οι διάφορες κυβερνήσεις. Τώρα, τέταρτη ερώτηση όντως ε, τα μικρά κράτη αντιμετωπίζουν προβλήματα να βρουν τους απαραίτητους πόρους σε τεχνολογικό και οικονομικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Το εξετάσαμε αυτό και εμείς πολύ προσεκτικά και δεν οφείλεται στο γεγονό ότι προερχόμαστε από μικρές χώρες, αλλά ε, επίσης το πώς οι μεγάλες χώρες υποστηρίζουν τις προσπάθειες αυτές είναι επίσης σημαντικό τα κράτη-μέλη, τα μεγάλα κράτη-μέλη δίσταζαν να, να ακολουθήσουν τις συστάσεις ε, της Κομισιό. Βέβαια, σε διμερές επίπεδο υπάρχει βοήθεια αν κάποιος τη ζητήσει. Και κάποιες μικρές χώρες, ε, χωρίς να τις αναφέρω βέβαια, να σας πω ότι είχαν ε, καλά αποτελέσματα όταν ζήτησαν τη βοήθεια των μεγαλύτερων χωρών. Επίσης μπορούν να βοηθήσουν και τη βοήθεια της ΕΝΙΖΑ. Τώρα, σε διμερές επίπεδο οι μεγάλες χώρες προσέφεραν υποστήριξη, όμως πολλές φορές τα κράτη-μέλη δεν αφιερώνουν ε, τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους και σε, δεν, δεν χρησιμοποιούν κάποιον υψηλά στην ιεραρχία όπως τα μικρότερα κράτη. Ούτως ή άλλως στις ε, ομάδες ε, για τη διαμόρφωση της πολιτικής εφόσον δεν είναι τα κατάλληλα άτομα παρόντα δεν μπορούν να ληφθούν και οι αποφάσεις. Θα ήθελα επίσης να το αναλύσω λίγο το θέμα περαιτέρω. Δεν είναι συχνές οι άμεσες επιθέσεις από χώρα σε χώρα γίνεται μέσω μιας άλλης χώρας η επίθεση που παίζει αυτή και αυτή η χώρα, η τρίτη χώρα είναι η, η ενδιάμεση χώρα. Τον Ιούλιο του 2010 οι Ηνωμένε Πολιτείε υπέστησαν μια επίθεση. Οι πέντε, πέντε σερβερς χρησιμοποιήθηκαν για αυτή την επίθεση. Μία από αυτές ήταν στην Αυστρία. Εάν όμως ε, η Γερμανία ας πούμε στην, ε, ε, είχε υποστεί αυτή την επίθεση και μία από τις πηγές επίθεσης ήταν η Αυστρία θα γινόταν μια φοβερή, φοβερή συζήτηση για το πώς μπορεί η Αυστρία να βοηθήσει μια χώρα εταίρων. Καταρχάς θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι τα νομικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει τα απαραίτητα νομικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε μια επίθεση την οποία δεν θα υποστούμε εμεί, αλλά θα την υποστεί μια άλλη χώρα. Και αν δεν ε, γίνει κάτι τέτοιο, οφείλω να ομολογήσω ότι θα είμαστε ιδιαίτερα ευάλωτοι, διότι θα κινδυνεύουμε να υποστούμε μια επίθεση από μια τρίτη χώρα που θα είναι μικρότερη από εμά. Για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα και οφείλεται σε δύο ε, παράγοντες. Ε, καταρχάς αφορά τους πολίτες και αφετέρου την, τις, τις υπηρεσίες προφοριών και κατασκοπίας. Και απέχουν πολύ το ένα σκέλος από το άλλο. Και για μια επίθεση δεν είναι αναγκαία το αρνητικό, διότι μια τράπεζα που δίνει πληροφορίες μπορεί να πει ότι υφιστάμεθα επίθεση στο λογισμικό και για την διάθεση πληροφοριών στους ε, κύβερνο-στρατιωτικούς ε, ε, θα υπήρχε η ανταπόκριση ότι πρέπει να ανταποκριθούμε. Είναι λοιπόν η ξεχωριστή δραστηριότητα, κάτι το οποίο μπορεί να είναι θετικό. Και σε σχέση με το πώς έχουν δημιουργηθεί στις ΕΠΑ αυτές οι δομές, είναι ενδιαφέρον. Στην Ευρώπη συμφωνούμε ότι αυτό δεν είναι μείζον θέμα για μας, διότι το στρατιωτικό σκέλος δεν θα έπρεπε συχνά να είναι ε, ο επικεφαλής στις ε, κυβερνοεπιθέσεις. Είναι αρμόδιοι στρατιωτικοί για τη δική τους ασφάλεια, για τη δική τους ε, κυβερνοάμυνα. Πρέπει να προφανώς να επιζητεί τη συνεργασία σε σχέση με άλλες χώρες, όμως σε σχέση με την επίθεση που θα δεχόταν μια χώρα είναι συντονιστικός ο ρόλος. Βλέπουμε ότι είναι ένα θέμα της χρήσης των βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με μια χώρα και γι' αυτό ίσως ε, αυτό που μπορώ να αναφέρω είναι δύο. Το κέντρο διαχείρισης κρίσεων στη Γαλλία που έχει ε, ε, καλές επιδόσεις ε, φαίνεται όμως ότι βρίσκεται υπό τον πριτανεύοντα ρόλο των ε, ε, στρατιωτικών αλλά και το κέντρο στην Γερμανία που θεωρώ ότι έχει μια θετική συνιστόσα βρίσκονται εκτός στρατιωτικού σκέλους και είναι, υπόσχονται να είναι πολύ πιο αποδοτική και αποτελεσματική και σε σχέση με τις λεπτομέρειες σε σχέση με άλλα κράτη το ε, ελβετικό πρότυπο είναι εκείνο το οποίο θα μπορούσε να ανταποκρίνεται σε ε, μεσαίου μεγέθους χώρες. Είναι ε, πολύ αποδοτικοί, έχουν το σκέλος στην πολιτική δράση που είναι αποτελεσματικό και που δίνει τη δυνατότητα η πολιτική ηγεσία να διαβουλεύεται. Έχουν όμως και μια ευρύτερη στρατιωτική βάση αυτό όμως ε, δεν ε, εμπλέκεται στις ε, καθημερινές δραστηριότητες, μόνο αν υπάρχει μια μεγαλύτερη κρίση εμπλέκεται αυτό το σκέλος. Επίσης, όσον αφορά για την κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να αναφερθώ στην προηγούμενη απάντηση που έδωσα. Δεν είναι η χρήση hackers για να χτυπήσουμε τους hackers αλλά η χρήση των δυνατοτήτων της κοινωνίας των πολιτών για να αυτοπροστατευτεί, να κάνει ό,τι είναι αναγκαίο ώστε να προστατευτεί έναντι άλλων πτυχών που αφορούν μη κρατικούς φορείς ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Να μπορέσουμε έτσι να ανταποκριθούμε σε σχέση με το σκέλος αυτών των δράσεων. Διότι στο τέλος τέλος τα στοιχεία από πλευράς ε, πληροφοριών αν υπάρχει ε, αποσαφήνιση των θεμάτων ε, κρατικής ή μη επίθεσης βλέπουμε ότι θα μπορούσε αυτό να ληφθεί υπόψη. Τώρα το ότι μη κρατικοί φορεί θα ε, επιζητούν οικονομικού χαρακτήρα πληροφορίες και ε, θα μπορούσαμε σε αυτό το επίπεδο να δραστηριοποιηθούμε. Κάποιε από τι επιθέσει που γίνονται είναι τόσο περίπλοκε και σύνθετε και είναι τόσο μυστικέ που δεν έχουν ποτέ καλυφθεί από τα μέσα ενημέρωση και μόνο από κρατικού φορεί ε, καλύπτονται. Όμω μπορούν κρατικοί φορεί να, δραστηριοποιούνται όταν υπάρχει ε, τέτοιου είδου επίθεση και ο στρατηγό Μάικο Χέιντεν, επικεφαλή ε, σε σχέση με τι δράσει για την CIA, οι δηλώσει του φυσικά εκφράζουν την αμερικανική τοποθέτηση ότι η κατασκοπία στην κυβερνοχώρου είναι μια κανονική δραστηριότητα. Αν προσπαθεί κάποιο να κλέψει τι δικέ μου πληροφορίε ε, και καταφέρει να τις κλέψει, τότε ε, εγώ φταίω και όχι εκείνος που τις έκλεψε, γιατί εγώ δεν μπόρεσα να αυτοπροστατευτώ. Μη κρατική όμως φορείς ε, από την άλλη πλευρά είναι ένας μεγαλύτερος κίνδυνος και υπάρχει και μια ε, ερώτηση που δίνει συνέχεια σε αυτή την πτυχή. Είναι επικίνδυνη επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κυβερνήσεις αυτοί οι μη κρατικοί φορείς και μπορούν να δράσουν και ανεξάρτητα. Δεν γνωρίζουμε αν ενεργούν για λογαριασμό τους υποκρατικό έλεγχο και τα δίκτυα κατασκοπίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες σε περίπτωση επίθεση. Όταν υπάρχει επίθεση από έναν μη κρατικό φορέα, πώς γνωρίζει, μπορεί να γνωρίζει κανείς, αν είναι η ενδεχόμενη κυβέρνηση που εμπλέκεται ή όχι, όταν έχουμε ένα μη κρατικό φορέα που μπορεί να δρά για λογαριασμό του ή έχουμε κάποιον που μπορεί να δρά για κάποιον τρίτο και χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για να... και ξεκινά μια κυβερνοεπίθεση. Αυτά είναι τα σενάρια για τα οποία γίνεται λόγο σήμερα και γι' αυτό ο πραγματικός κυβερνοπόλεμος μπορεί και τυχαία να ε, εκραγεί συγκυριακά. Τώρα, η αποφυγή των ε, ε, διπλοεπικαλύψεων και αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ε, δούμε το ότι ο κάθε ένας κάνει ξεχωριστό, έχει ξεχωριστό έργο. Το ΝΑΤΟ για παράδειγμα σε σχέση με την CIP και όσον αφορά τις, τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχει το ΝΑΤΟ στην υπηρεσία του αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομίζω μεγάλος κίνδυνος δίπλο και επειδή ίσως θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το, τόση μεγάλη η εμβέλεια, η, αναλογία των δράσεων του ε, ΝΑΤΟ ως προς αυτό. Και τώρα για τα υπόλοιπα ε, εντάχει, για την Κίνα και την Ρωσία σε σχέση με το αν είναι ή όχι αντίπαλοι ή εχθροί. Υπάρχουν εδώ κοινά στοιχεία και μας απασχολούν σε σχέση με την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος για παράδειγμα όσον αφορά την Ρωσία θα πρέπει εφόσον υπάρχει έτοιμα να τους υποστηρίζουμε φυσικά και να τους συνδράμουμε για την Κίνα σε σχέση με τον, ε, την δυνατότητα εξυγχρονισμού μπορούμε να ε, παράσχουμε υπηρεσίες. Δεν μπορώ να σχολιάσω οποιασδήποτε δράσεις από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Εν τέλει νομίζω ότι αν η ΕΠΑ μια και έχουν ενεργό ενδιαφέρον να συνεχίσουν ε, να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να αποτρέψουν επιθέσεις ε, αυτό είναι σημαντικό για το κόστος υπάρχουν κάποιες μελέτες που έχουν ε, συνταχθεί μπορείτε διμερώς να έρθετε σε επαφή μαζί μου για αυτά τα στοιχεία υπάρχει και η επίπτωση μελετών για τις ε, ε, επιπτώσεις των κυβερνοεπιθέσεων στη ΣΥΠΑ. Έχει γίνει και μια μελέτη για την Ελβετία. Δεν υπάρχει μια μελέτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να γινόταν σε σχέση με τα κόστη. Πρόληψη, μάλιστα. Η πρόληψη... Δεν μπορώ να δώσω βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη Ουσιαστικά πρόκειται για μέτρα για την κυβερνοασφάλεια που θα μπορούσαν να είναι η καλύτερη πρόληψη. Αφορά και τους ιδιώτες, ποια ηλεκτρονικά μηνύματα ανοίγουν και πώς προσεγγίζουν αυτό το σκέλος το, της επικοινωνίας, γιατί και εκεί μπορεί να υπάρχουν ε, τέτοιου είδους ενδεχόμενα μιας ε, ε, προσβολής. Αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο ακαδημαϊκά σε θεωρητικό επίπεδο έχουμε συζητήσει. Από τη μία πλευρά θα πρέπει να μπορεί η άμυνα να είναι εφάμιλη καλύτερη από την επίθεση. Σε σχέση με τις μελλοντικές προοπτικές δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει. Όλα αυτά δείχνουν πόσο περίπλοκα είναι τα πλαίσια. Πρέπει να εξειδικεύσουμε τις μελέτες μας και όταν έχουμε καλύψει κάθε εξειδικευμένη λεπτομέρεια τότε θα είμαστε ίσως καλύτερα προετοιμασμένοι. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι η ε, τη δεκαετία του 1980 ήταν οι πρώτες ε, επιθέσεις hardware attack είχαμε ε, σε σχέση με, την, με ένα σενάριο επίθεσης που θα ήταν καταστροφικό γίνονται όμως σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων της ίδιας που υπάρχουν chips ημιαγωγή και υπάρχει και η χρήση ε, των θεμάτων κώδικα από τις ε, ε, υπηρεσίες. Είναι αδύνατο να υπάρξει απόλυτη προστασία έναντι τέτοιου είδους επιθέσεων. Είναι πάρα πολύ σοβαρά ενδεχόμενα. Και όταν κάνουμε λόγο για χώρες σε κυβερνοσύγκρουση είναι Κάτι το οποίο ποτέ εκεί δεν μπορεί να εμπλέκει τους ε, ε, εκτός κρατικούς φορείς. Πάντα θα είναι κάποια κράτη τα οποία θα εμπλέκονται σε αυτή την εμβέλεια της σύγκρουσης. Νομίζω ο Αλέξανδρος έδωσε μια πολύ καλή επισκόπηση για την λειτουργική ανταπόκριση για την περισσότερο στρατιωτική θα έλεγα το συνιστόσα αυτού του θέματος. Ως ε, υπάλληλος, κυβερνητική υπάλληλος ε, προσεγγίζοντας ε, τα θέματα της ε, κυβερνοπροστασίας υποκυβερνητικό πρίσμα. Ίσως θα μπορούσα να κατηγοριοποιήσω τις ερωτήσεις σας σε ομάδες για να απαντήσω πιο αποτελεσματικά. Πρώτον, από πολλές ερωτήσεις αποδεικνύεται ότι υπάρχει κάποια σύγχυση. Ποιο είναι εκείνο ο οποίο θα απαντά από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα υπουργό άμυνα, ε, υπουργό εσωτερικών, ε, η ε, κοινότητα για την, τα θέματα ασφάλεια. Όταν κάναμε αυτή τη μελέτη για την διάρκεια, α το πω έτσι, για εξάμεινη προοπτική, τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να πει κανείς ε, για μια τέτοια ανταπόκριση. Η απάντηση είναι ότι εσείς θα πρέπει να απαντήσετε επί τόπου άμεσα και για, επειδή πρέπει να προστατέψετε τα δίκτυά σας και δεν είναι δυνατόν να εγκαταλείψετε την προστασία της χώρας σας. Δεν είναι λοιπόν το σημαντικό ποιος θα απαντήσει, αλλά να υπάρξει απάντηση. Κάποιος να, ενεργοποιήσει αυτή την απάντηση. Και υπό συμβατικούς όρους μέσα στο κυβερνοπλαίσιο αυτό το θέμα δεν έχει τέτοια μεγάλη σημασία. Αν δει κανείς την εξέλιξη των συγκρούσεων και από την εξέλιξη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που είχαμε μετά από αυτόν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την τα βομβαρδιστικά και τις αεροπορίες ε, που ε, ε, οργάνωναν πλήγματα η διαμόρφωση των πληγμάτων και της σύγκρουσης στο μέλλον μεταβάλλεται. Ο ρόλος και η παραδοσιακή σημασία των στρατιωτικών σε μεγάλη κλίμακα τέτοιες εχθροπραξίες θα είναι μικρός. Λυπούμε που πρέπει να το πω αυτό. Θα έχουν κάποιο ρόλο αλλά όχι τόσο μεγάλο ρόλο. Για να ανταποκριθείτε σε τέτοιου είδους κυβερνοεπιθέσεις θα πρέπει η ευρύτερη κοινωνία να μπορεί να ανταποκριθεί και να προστατευτεί διότι όλες οι υπηρεσίες σε μια τέτοια ευρύτερη κυβερνοεπίθεση θα πληγούν. Έχουμε τις εταιρείε, έχουμε τις υποδομές που υποστηρίζουν τις εταιρείε αυτές, την τροφοδότηση των υποδομών. Είναι ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη αλυσίδα. Οι στρατιωτικοί δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, έχουμε υπεύθυνους που βρίσκονται σε ε, βάσεις ηλεκτρονικών δεδομένων και που πρέπει να απαντήσουν όμως ε, σε μια τέτοια επίθεση. Όμως ε, είναι πολύ ευρύτερο το φάσμα και μια κυβερνοεπίθεση είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μια αποσύνδεση. Όμως θα πρέπει κανείς να δει ότι πρέπει να αποφευθεί η ε, μεγαλύτερη ζημιά. Όλη αυτή η ε, διαπλοκή αυτών των θεμάτων είναι κάτι που πρέπει με καινοτομία, με καινοτόμο τρόπο να μας κάνει να δραστηριοποιηθούμε ώστε να εξεύρουμε μεθόδους και μηχανισμούς πολιτικής αντίδρασης στο εθνικό επίπεδο, στο κρατικό επίπεδο και μετά από αυτό στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι στο τοπικό επίπεδο πρέπει να υπάρχει η απάντηση σε μια κυβερνοεπίθεση. Δεν έχει νόημα να περιμένουμε να δοθούν κάποιες εντολές ή κάποιες δράσεις να αναλυφθούν πρώτα στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι βέβαια σημαντικό να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως πρέπει σε τοπικό επίπεδο να αντιδράσει κανείς άμεσα αν υπάρξει πλήγμα. Γι' αυτό όλα αυτά τα συστήματα στα διαφορετικά κράτη-μέλη όπου υπάρχουν θέματα κέριων υποδομών και επαΐοντες εμπλέκονται στην διαχείριση στο κρατικό επίπεδο σε σχέση με αυτές τις υποδομές το ίδιο ε, ισχύει και για την Εστονία αυτή είναι η σωστή μεθοδολογία ανταπο, αντίδρασης σε αυτού του είδους ε, τις επιθέσεις συμφωνώ με την παρατήρηση ότι η πρόληψη είναι πιο αποτελεσματική από την ε, ε, το, το πλήγμα ε, στην, μετά την επίθεση, μετά την εκδηλωμένη επίθεση. Όμως όλα εξαρτώνται από το πώς θα μπορέσει να δράσει κανείς. Αν δεν είναι σημαντικές οι επιπτώσεις ε, δεν έχει νόημα να ξεκινήσει μια εθνική αντίδραση. Αν δύο τράπεζες έχουν υποστεί επίθεση σε μια τράπεζα, αρνητικό είναι αυτό βέβαια για αυτές τις δύο τράπεζες που έχουν υποστεί τέτοιες επιθέσεις. Αν όμως χιλιάδες επιθέσεις αποτελούν στόχο επιθέσεων, τότε πρέπει να ξεκινήσει μια εθνική ανταπόκριση, μια εθνική ε, αντίδραση. Και μετά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναλογικά το ίδιο. Εδώ θα μπορούσαμε ίσως ε, να δούμε λιγότερη ας το πω έτσι ε, παρενόχληση ε, όσον αφορά το, τις μελλοντικές δράσεις μεγαλύτερη αντιμετώπιση πιέσεων ε, ή πληγμάτων όπως στην Εστονία με ασύμετρες δράσεις ίσως κάποιο γειτονικό κράτος ήθελε ή θέλει να δείξει στη μικρή Εστονία ότι οποτεδήποτε επιθυμούμε μπορούμε να σας διαλύσουμε αυτού του είδους ας το πω έτσι χρήσης, η χρήση μη συμμετρικών μέτρων ή ασύμμετρης ε, ε, αναλογίας δύναμης είναι ε, στοιχείο το οποίο εμπεριέχεται εδώ. Πολλοί κρύβουν επιθέσεις, μπορούν και κρύβονται πίσω από κάποιους άλλους όταν υπάρχει επίθεση έναντι στόχου. Για παράδειγμα αυτό έγινε στην Γεωργία στο παρελθόν Όλα αυτά θα γίνονται πιο αυξημένα στο μέλλον και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ενδυνάμωση της ε, διεθνούς ε, νομικής πτυχής ε, όσον αφορά την αντίδραση. Όταν υπάρχει η αποσαφήνιση της εθνικής ευθύνης από πλευράς ενός κράτους μέλους μπορεί να υπάρξει νομική, ας το πω έτσι, αντίδραση σε σχέση με το διεθνές δίκαιο ή με, τον, με διεθνή δικαστήρια που μπορούν να εμπλακούν. Αυτό είναι μια σημαντική πτυχή όσον αφορά το μέλλον. Και εδώ θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε να διαδραματίσει πολύ πιο ενεργό ρόλο σε αυτέ τι συζητήσεις. Όσον αφορά όμω την αναλογία, η αναλογικότητα, πώς αντιδρά κανείς, θα έπρεπε με αναλογικό τρόπο, με αναλογικότητα να μπορεί κανεί να αντιδρά. Επίθεση εναντίον μια εταιρεία από κυβερνοεγκληματίε, η αντίδραση θα είναι η επιβολή του νόμου, η προσαγωγή στα δικαστήρια για τις περισσότερες ε, επιθέσεις ε, υπάρχει κάποιο κίνητρο σε σχέση με αυτές τις επιθέσεις. Υπάρχει όμως ε, και κατασκοπία και βιομηχανική κατασκοπία και αν κάνει κανείς τον λόγο, κάνει λόγο για το κόστος για τις οικονομίες μας είναι ένα είδος κυβερνοεγκλήματος που είναι πάρα πολύ δαπανηρό. Συνεπάγεται πολύ μεγάλα κόστη. Ακόμα και οι ε, εγκληματίες του κυβερνοχώρου οι οποίοι έχουν ε, εξειδικευθεί και ε, δρούν συνενωμένα είναι πολύ επικίνδυνοι. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν η λήψη υπόψη του κόστους αυτού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως οι συνάδελφοι από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ασχοληθεί με αυτό. Οι εταιρείε όμως δεν αποκαλύπτουν τα ποσά. Τι έχουν απολέσει δηλαδή δηλαδή. Και αυτό είναι ουσιαστικό στοιχείο. Όταν κάνει κανεί λόγο για στατιστικά στοιχεία κυβερνοεγκληματικών περιπτώσεων, δεν υπάρχουν ε, τα σωστά αριθμητικά μεγέθη, τα σωστά στοιχεία για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τι περιπτώσει. Πόσα εγκλήματα, πόσα πλήγματα υπήρξαν, ποια ήταν η συνολική ζημιά από τέτοιου είδου επιθέσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα όσο έχει σήμερα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, να πούμε για τα μέτρα που έχει ε, υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλά έχει επενδύσει σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου και την επιβολή του νόμου και του δυναμικού της εφαρμογής του νόμου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το σκέλος εξελίσσονται οι προσπάθειες και περισσότερα κονδύλια θα πρέπει σαφώς να ε, κατανεμηθούν σε αυτές τις δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο. Αυτό το οποίο τώρα έχουμε και διακυβεύεται είναι θέματα διακυβέρνησης ε, της, ε, στον κυβερνοχώρο. Δεν είναι μόνο θέματα ασφάλειας, ε, είναι το θέμα της διακυβέρνησης του κυβερνοχώρου. Πώς είναι κανείς σε θέση είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο εταιρεία, είτε σε οργανωτικό επίπεδο να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει λογοδοσία, διακυβέρνηση χρηστή και ορθή και σωστή αντίδραση ή ανταπόκριση σε αναλογικό επίπεδο σε οποιαδήποτε ενδεχόμενα. Είναι ένα θέμα διοργανωτικό. Είναι μια νέα πορεία. Πορευόμαστε και διανύουμε παρθένο έδαφος, αλλά μπορούμε να δούμε την πτυχή της συνιστώσας των κρατών μελών, τις ε, πτυχές της διοργάνωσης ε, εταιρικά ή επιχειρησιακά. Το θέμα μεγάλων και μικρών κρατών μελών, αυτό είναι τεχνητή, τεχνητός διαχωρισμός. Στον κυβερνοχώρο όλοι είμαστε ίσοι. Και αυτό ίσω είναι ένα μείζον πρόβλημα. Ίσως οι μεγαλύτερε χώρε έχουν μεγαλύτερο δυναμικό να διαθέτουν κονδύλια, αλλά ταυτόχρονα είναι και πιο ευάλωτε οι μεγαλύτερε χώρε, επειδή μπορούν πολλαπλά να αποτελέσουν στόχο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν άσχετα από το μεγάλο ο μικρό, πρέπει, είναι αληθεύει βέβαια ότι οι μικροί πρέπει να αναλώνουν, να, να, να δαπανούν ε, περισσότερα κονδύλια για να διασφαλιστεί η ελάχιστη ικανότητα από πλευρά του ε, να μπορούν να αντιδράσουν. Για το θέμα που αφορά το ΝΑΤΟ, που αναφέρθηκε και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται προ στην ορθή πορεία θα έλεγα. Μια στρατιωτική οργάνωση είναι το ΝΑΤΟ που προσπαθεί πρώτα απ' όλα να προστατεύσει τα δικά του συστήματα και τα τηλεπικοινωνικά του συστήματα σε περίπτωση κρίσεων ε, και διοργανωτικά να μπορέσει να προστατευτεί. Είναι στρατιωτικού χαρακτήρα. Δεν θα περάσει στο πολιτικό σκέλος ε, ε, το ΝΑΤΟ Ωστόσο, το άρθρο 5 επιλύεται, ανταποκρίνεται τον ΝΑΤΟ. Μπορεί να απαντήσει το ΝΑΤΟ και να ενεργοποιηθεί. Μπορεί δυνητικά αλλά δεν λέει και δεν αποσαφηνίζει πώς και με πιο ακριβώς τρόπο. Και εδώ υπάρχει και το θέμα της ελαστικότητας ε, ε, της ε, ανταπόδοσης ή της ανταπάντησης. Θα πρέπει λοιπόν να, το, να υπάρχει το ενδεχόμενο ή της πολιτικής ή της στρατιωτικής ή της συλλογικής απάντησης από πλευράς του ΝΑΤΟ όταν και αν χρειαστεί ο επιμερισμός του έργου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ακόμα στο πολιτικό σκέλος αυτού του σκηνικού, το ΝΑΤΟ στο, πιο, στο στρατιωτικό, όμως ταυτόχρονα μπορούν να συνδέσουν και να συνενώσουν τις ε, δυνάμεις τους, να ανταλλάξουν πληροφορίες ή έγκαιρα ε, μέσω συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν μέσα από αυτή τη συνεργασία. Πρέπει να διασφαλιστεί αυτή η συνεργασία. Πρέπει να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός και στο εθνικό αλλά και στο πανενωσιακό ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε ευθύ στο δεύτερο πάνελ με τον κύριο Βιλαλόγκα και την Επιτροπή. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που καλέσατε την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής δράση να συμμετέχει στην παρουσίαση της μελέτης αυτής και στη συζήτηση για το κυβερνό και την κυβερνό ασφάλεια. Είναι και μεγάλη χαρά μου αλλά και μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μιλήσω στην Υποεπιτροπή ε, του Κοινοβουλίου για την ε, ασφάλεια και την άμυνα σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια και το έγκλημα. Ελπίζω όταν τελειώσω την ε, παρουσίασή μου να μην ε, σας μείνει η εντύπωση ότι δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό στο πλαίσιο τη και πάει ίσω αυτό στο παρελθόν να γινόταν, αλλά μέχρι τώρα ε, βλέπουμε ότι έχουν ληφθεί πρωτοβουλίε και έχουν υπάρξει εξελίξει και πολύ πρόσφατε που έχουν βάλει πολύ ψηλά στην ατζέντα τη ΕΙΕΔ τα θέματα τη κυβερνοασφάλεια. Λέγομαι Χωακίν Βιλελόγκα και είμαι επικεφαλή του τμήματο για την ασφάλεια, στην ΕΙΕΔ. Το τμήμα αυτό ε, της πολιτικής ασφάλειας προσπαθεί να εφαρμόσει την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργαζόμαστε βέβαια και με άλλες ε, διευθύνσεις. Προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε τις προτεραιότητές μας σε όλο το έργο της ΕΕΔ με κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Πολιτικό διάλογο με τις χώρες για θέματα ασφάλειας έως στρατηγικό προγραμματισμό μέσα συνεργασίας, μέσα ενίσχυσης και πολλά μέτρα για τα οποία είναι αρμόδια η υπηρεσία μας, το τμήμα μας. Βέβαια, συνεργαζόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το Συμβούλιο αλλά και με τα κράτη-μέλη και βέβαια όπως σήμερα και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα της διάστασης της εξωτερικής ασφάλειας και της εσωτερικής ασφάλειας. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διασύνδεση μεταξύ εξωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Η κυβερνασφάλεια και το κυβερνοέκλημα νομίζω είναι το πιο απτό παράδειγμα διότι τίθεται θέμα ασφάλειας όχι μόνο για του ιδιώτες αλλά και για δημόσιους ιδιωτικούς οργανισμούς, για ολόκληρα κράτη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα της ασφάλειας ε, και αυξάνεται η σημασία του γιατί υπάρχει όλο και μεγαλύτερη διασύνδεση. Νομίζω ότι δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε σήμερα ότι χωρί κυβερνοασφάλεια δεν υπάρχει ασφάλεια. Οι κυβερνοεπιθέσει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορου ε, στόχου, εγκληματικού ε, μεταξύ αυτών και βέβαια η συνολική ζημία είναι εκατοντάδες δις ευρώ. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν επίσης για κατασκοπία, κατά κυβερνήσεων, κατά στρατιωτικών ε, ε, υποδομών ή για πολιτικό εξαναγκασμό, εκφοβισμό, να επηρεάσουν σχέσεις μεταξύ κρατών ή μπορούν να στηρίξουν διασυνορικές στρατιωτικές επιθέσεις. Είχαμε πρόσφατα το επεισόδιο Stoxnet και έδειξε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, το κυβερνέτημα και για ε, το σαμποτάζ, τη δολιοφθορά κατά ε, κυβερνητικών ε, υποδομών. Το 2008 η κυβερνοασφάλεια θεωρείται προτεραιότητα τη εξωτερική σα πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζεται η οικονομική και η στρατιωτική σημασία και ζητείται μια μεγαλύτερη συνεργασία και συντονισμό. Οι κυβερνοαπειλέ επίση και στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης και στην εσωτερική ε, πολιτική και τα σχετικά έγγραφα λαμβάνουν και μεγαλύτερη σημασία. Σε ό,τι αφορά το ρόλο της ΕΙΕΔ, θεωρείται ότι αυτό το πρόβλημα που είναι παγκόσμιο μπορεί να το πιστεί μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή με συνεργασία. Θα σας δώσω μόνο δύο παραδείγματα. Με τις, ε, με τις είπα, όπως ξέρετε, σήμερα και το 2010 σε Σύνοδο Κορυφή συστήθηκε, συστάθηκε μια ομάδα εργασίας για την κυβερνοασφάλεια μετά από τις δηλώσεις ε, της Συνόδου Κορυφής του 2009 που αναγνωρίζει την στρατηγική σημασία για την δυνάμωση του διαλόγου ασφαλείας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΕ και φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι από την Κομισιό θα σας ενημερώσουν ε, για τις εργασίες αυτής ε, της ομάδας. Επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι στις 16 Μαΐου, δηλαδή λιγότερο από ένα μήνα πριν, οι ΙΠΑ δημοσίευσαν την εσωτερική στρατηγική για τον κυβερνοχώρο και το έγγραφο αυτό τονίζει την ανάγκη διεθνού συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή και αναφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση ω εταίρο για αυτή τη συνεργασία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Ινδία στα περιθώρια της Συνόδου Κορυφής μεταξύ των δύο πλευρών ε, το Δεκέμβριο συμφώνησαν οι τεχνικοί σύμβουλοι να ε, ε, διευρύνουν τη συνεργασία τους και στον τομέα της ασφάλειας. Και η ΕΕ σε αυτό το πλαίσιο έχει καλέσει σε εμπειρογνώμονες να μας ενημερώσουν για, τους, για τις διάφορες εξελίξεις και βέβαια συνεργαζόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρξει και ένα σεμινάριο από, ένα κοινό κέντρο, από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Επίσης, συνεργασία με τον ΝΑΤΟ για τα θέματα της κυβερνοασφάλειας. Ξέρετε ότι υπάρχει το νέο στρατηγικό δόγμα που, ε, εγκρίθηκε στη Λισαβόνα τον νοέμβριο. Μεταξύ αυτών η κυβερνοαπειλή είναι πάρα πολύ ψηλά στην ε, ε, ατζέντα Υπάρχει ε, η πρόταση για την κυβερνοασφάλεια και τη σχετική πολιτική που μάλλον τον Ιούνιο θα εγκριθεί. Υπάρχουν δραστηριότητε κοινέ, ανταλλάσσουν πληροφορίε, είμαστε σε επαφή και προσπαθούμε να προωθήσουμε την αλληλοσυμπληρωματικότητα. Επίση, η κυρία Άστον στι συζητήσει που έχει με τον ε, κύριο Ράσμουσεν, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αναφέρει ω προτεραιότητα τα θέματα τη κυβερνοασφάλεια. Για πρώτη φορά, επίση, βλέπουμε το ενδεχόμενο το κυβερνοέγκλημα και η κυβερνοασφάλεια να είναι μία από τις νέες βασικές προτεραιότητες της μακροπρόθεσμης συνιστώσας του μέσου για τη σταθερότητα. Και επεξεργόμαστε τη στρατηγική που θα υποβάλουμε μάλλον στα κράτη-μέλη και την συγκεκριμένη επιτροπή τις προσεχείς εβδομάδες. Θέλουμε να στηρίξουμε την ανθεκτικότητα και την αντοχή και τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και των εταίρων μα και των γειτόνων μα για να μπορούν όλοι να αντιδρούν γρήγορα σε κυβερνοεπιθέσει και να εντοπίζουν και να διώκουν του εγκληματίε ε, του κυβερνοχώρου. Θα πρέπει να υπάρχουν ομάδε αντιμετώπιση επιγόντων περιστατικών, θα πρέπει να θεσπιστούν ε, νομικά πλαίσια και να υπάρξει και διεθνή συνεργασία με βάση τα πρότυπα της Σύμβασης της Βουδαπέστης. Θα ήθελα επίσης για να σας ενημερώσω για το PSE Υπάρχει εντολή για θέματα εξωτερικής ασφάλειας και ήδη έχει συζητηθεί το θέμα της κυβερνοασφάλειας σε αυτό το πλαίσιο. Και σε αυτό που θα σας ενδιαφέρει ίσως είναι ότι την 1η Ιουνίου, δηλαδή ε, πριν από λίγες ημέρες, έγινε μια κοινή συνάντηση με την ΚΟΣΗ, εσωτερική ασφάλεια, και τέσσερα ήταν τα θέματα στην μέση διάταξη μόνο. Ένα από αυτά ήταν ακριβώς πώς μπορεί να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής διάσταση τη κυβερνοασφάλειας. Βλέπετε λοιπόν ότι ο κυβερνοχώρος είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για την ΕΕ και όλες οι υπηρεσίες συνεργάζονται μεταξύ τους. Αλλά συνεργαζόμαστε και με τους διεθνούς μας εταίρους. Ε, τώρα, έχουμε και με το στρατιωτικό μας προσωπικό, έχουμε και την, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας βέβαια που δραστηριοποιείται στο θέμα του κυβερνοχώρου, το στρατιωτικό προσωπικό εδώ και τρία χρόνια εξετάζει αυτά τα θέματα. Είχαμε και το σχέδιο ανάπτυξη δυνατοτήτων του 2009. Θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να ευνοήσουμε και τα εσωτερικά στρατιωτικά ε, δίκτυα εντό δηλαδή Ένωση για να παρέχουν, επικοινωνία, να παρέχουν ανακοινώσει, αλλά και πώ μπορούμε να προωθήσουμε και κάποια μέτρα μετριασμού των απειλών. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ο Οργανισμός Άμυνας έχει μια ομάδα για την κυβερνοασφάλεια, συμμετέχει και το στρατιωτικό προσωπικό, το τμήμα πολιτικής, ε, το δικό μας, αλλά και το ένιζα. Επίσης, είμαστε και ένα σημείο επαφή ένα εστιακό σημείο διότι είναι πολύ πολύπλοκοι οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι δύσκολο πολλές φορές να καταλάβουμε τι ε, είναι η αρμοδιότητα ποιου. Και πολλές φορές υπάρχουν ζητήματα τα οποία τα ε, παραπέμπουμε στους αρμόδιους και στα κράτη-μέλη και στην Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση διεθνή βήματα συζήτησης, κυβερνοασφάλεια και κυβερνοέγκλημα είναι αντικείμενο 30 ε, οργανισμών, ο ΟΣΑ, ο ΑΣΕ, περιφερειακές οργανώσεις, ε, οργάνωση Αμερικανών Πολιτειών κτλ. Και στην Κουαλά Λουμπούρ, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Φόρουμ της ΑΣΕΑΝ, επίσης ήμασταν εκεί για να συζητήσουμε τα θέματα της ασφάλειας. Επίσης, για τις διεθνείς ε, προδιαγραφές και πρότυπα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση αυτό τον καιρό. Υπάρχει και η διεθνή στρατηγική των ήπα για αυτά τα πρότυπα, πρόσφατα εγκρίθηκε. Και ο Υπουργό Εξωτερικών ε, της Αγγλίας Χέιγκ και ο κύριος Σαρκοζή ε, έκαναν σχετικές δηλώσεις στην Τοβίλτε ε, στο, το Μάιο. Και βέβαια θα πρέπει να προετοιμάσουμε την θέσεις μας για την διακυβέρνηση και την κυβερνοασφάλεια. Τα κράτη-μέλη έχουν, ασφάλεια, έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία στα θέματα τη κυβερνοασφάλειας. Υπάρχουν ε, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία που έχουν δημοσιεύσει πρόσφατα τις στρατηγικές εσωτερική ασφάλεια. πρέπει και εμεί να βασιστούμε στην εθνική εμπειρογνωμοσύνη για να αναπτύξουμε τι δικέ μα προτάσει, όπω είναι παραδείγματο χάρη του μέσου σταθερότητα. Επίση και με την Κομισιόν συνεργαζόμαστε, με τη ΔΕΛΤΑ ΕΜΣΟ, με τη ΔΕΛΤΑ HOME και με την ΔΕΛΤΑ Enterprise που κάνει σημαντική έρευνα σε αυτό το τομέα. Θέλουμε να υπάρχει στενό συντονισμό των δραστηριοτήτων μα. Πρόσφατα υπάρχει και μια διαπηρεσιακή υπηρεσία που συστάθηκε για την κυβερνοασφάλεια και το κυβερνό έγκλημα. Στις 6 Ιουνίου ε, συνήλθε για πρώτη φορά σε επίπεδο γενικών γραμματέων η ομάδα αυτή και ο κ. και ο Ανοπλωτή Γενικό Γραμματέα Υγεία, συμμετείχε σε αυτή την συνάντηση. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πρωτοβουλίε, υπάρχουν σημαντικέ εξελίξει ε, που ε, βάζουν την κυβερνοασφάλεια σε πολύ, ψηλό, σε πολύ ψηλή θέση στην ατζέντα τη ΕΙΕΔ. Όπω σα είπα, όπως βλέπετε κάποιες από τις συστάσεις ήδη ακούστηκαν από τους προλαλήσαντες ε, και ήδη γίνονται πραγματικότητα. Και θα ήθελα να σημειώσω και ε, τις άλλες βέβαια ε, συστάσεις και τα άλλα θέματα που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια και, την, και το κυβερνοέγκλημα. Θα πρέπει να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τα είπα πολύ γρήγορα γιατί δεν υπάρχει χρόνος και θέλω ε, να μιλήσει και η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριος ε, σέρβιτε τώρα. Good morning, Καλημέρα σας. Έχω να κάνω μία παρουσίαση, αλλά μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, δεν θα την παρουσιάσω. Το είχαν κάποιο την βάλει στην αίθουσα. Ε, το όνομά μου είναι Σερβίδα και είμαι ε, εκπρόσωπος της ε, Γενικής διεύθυνση για την Κοινωνία της προφορικής και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Θα ήθελα να κάνω μία παρουσίαση σύντομη για το πού βρισκόμαστε και ποιες είναι οι πράξεις που υιοθετήθηκαν από την Κομισιόν πρόσφατα και τελευταία τον Μάρτιο του 2011 όσον αφορά την ε, ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία των ευαίσθητων ε, πληροφοριών. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να δούμε ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά την πολιτική της κυβερνοασφάλειας στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλές πτυχές τις οποίες έχουμε εξετάσει. Καταρχάς βλέπουμε ποια είναι η απάντηση των, των πολιτών στα θέματα ε, διαταραχής του κυβερνοχώρου και Ε, πολλά από τα θέματα αυτά συζητήθηκαν και σήμερα το πρωί, ποιες είναι τα, είναι τα αποτελέσματα των επιθέσεων. Επειδή το βλέπουμε από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά της πρόληψης, ε, θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να υιοθετηθεί, τι θα πρέπει να εφαρμοστεί έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την δυνατότητα όχι μόνο να εντοπίσουμε ή να μετριάσουμε, αλλά να απαντήσουμε και να καλύψουμε πλήρως ε, κάποιες ε, επιθέσεις που μπορεί να διαταράξουν τον οικονομικό μας, ε, τον κοινωνικό μας χώρο. Ε, ούτως ή άλλως η διαταραχή, αν θέλετε, στην ζωή των πολιτών ή στον, οικονομική μας, στον οικονομικό μας χώρο ή στην, στον τομέα της διακυβέρνησης είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, ούτως ή άλλως ε, εδώ υπάρχουν, η απάντηση που να δώσουν οι πολίτες ή ο κυβερνητικό χώρος. Γι' αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε ε, την κουλτούρα της ασφάλειας, της καθημερινής ασφάλειας. Αυτό είναι εύκολο να το λέμε, αλλά δύσκολο να το κάνουμε εκτός και αν δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, αν θέλετε, στα θέματα της κυβερνοασφάλειας που να στηρίζεται στην διαχείριση του κινδύνου διαχείριση του κινδύνου το καν, την κάνουμε στον φορολογικό, στο δημοσιονομικό τομέα χάρη. Θα πρέπει να αυτή τη διαχείριση να την ε, διευρύνουμε και στον κυβερνοχώρο. Διότι η διαχείριση του κινδύνου είναι κάτι το οποίο όλοι μπορούν να καταλάβουν και πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν να παίξουν έναν ρόλο όλοι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι πρέπει να προστατεύσουμε, που είναι οι αξίες μας, τα χρήματά μας, αλλά τα, θα πρέπει να δούμε και ποια είναι τα εργαλεία, ποια είναι τα πιθανά εργαλεία τα οποία δεν πρέπει να τα αφήσουμε στα χέρια αυτών που μπορεί να έχουν εγκληματικές προθέσεις και μπορούν να διαπράξουν ε, τις επιθέσεις αυτές. Όλα αυτά ακούστηκαν και ε, προφανώς δεν μπορούμε να τα λύσουμε μέσα σε μια μέρα. Όμως οι αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα θα είναι σημαντικές για τα επόμενα 5 ή 10 χρόνια. Και αυτό γιατί, διότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις τεχνολογικές εξελίξεις ε, για τον, ε, ας πούμε, βλέπουμε πώς ε, ε, οι τηλεπικοινωνίες και η κινητή τηλεφωνία ε, ε, παρεμβαίνει στην, στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι έτοιμη να προωθήσει τις δικές της αρχές, τις δικές της αξίες και τις προτεραιότητες που θα ε, προωθηθούν σε διεθνές επίπεδο έτσι ώστε να διατηρήσουμε το ψηφιακό περιβάλλον ανοιχτό ε, ε, ποικίλο, διότι ούτω ή άλλω να υπάρχει μια τέτοια ποικιλία είναι καλό, ε, να υπάρχει μια διαλειτουργικότητα και αυτή είναι πολύτιμη, διότι υπάρχουν, όπως ακούσαμε, κράτη τα οποία βάζουν εμπόδια στο ίντερνετ και αυτός δεν είναι ένας καλός τρόπος για να αναπτύξουμε αυτό το περιβάλλον εάν θέλουμε το περιβάλλον αυτό να είναι ένας παράγοντας προώθησης και ανάπτυξης σε οικονομικό, κοινωνικό ε, και τεχνολογικό επίπεδο. Όμως θα πρέπει να ξεπεράσουμε το ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε σε μια διεθνή συνεργασία και ο συνάδελφος ε, από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων ε, τόνισε τον περίπλοκο χαρακτήρα της συζήτησης σε διεθνές επίπεδο. Τώρα, λίγα λόγια για το ποιες είναι οι πολιτικές μας, ποια είναι τα, αποτελέσματα, επιτεύγματα και ποιες είναι οι επόμενα, τα επόμενα βήματα. Το πρώτο βήμα είναι η ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη που είναι η βασική πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου Κρούσο, που είναι υπεύθυνο για την ε, κοινωνία της πληροφορικής και τις υπηρεσίες ε, για την ε, πολιτική δημιουργία των κρίσιμων αν θέλετε υποδομών Ούτως ή άλλως αυτό το οποίο θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να εξάγουμε συμπεράσματα από τα μέτρα τα οποία έχουν υιοθετηθεί μέχρι στιγμής. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες θα έλεγα για το πώς ε, τα διάφορα σενάρια απειλής εξελίσσονται. Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε την δυνατότητα ε, των ε, επιθέσεων στον κυβερνοχώρο να οδηγήσουν και σε φυσικές καταστροφές ε, δεν έχουμε δει τις συνέπειες ε, ε, τέτοιου συνέπειες των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο αλλά υπάρχουν συνέπειες σε, στον τομέα των, της ενέργειας, των μεταφορών ας πούμε η σημασία ενός remote control θα πρέπει να εξετάσουμε διάφορα σενάρια για, τις, για να δούμε ποια είναι τα ευάλωτα σημεία μας και το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες ε, επιθέσεις. Επίσης, ο στόχος αυτής της δήλωσης πολιτικής μας είναι να τονίσουμε ότι δεν ε, αρκεί μία ευρωπαϊκή προσέγγιση μόνο. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε ε, μια συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον κρίσιμο τομέα. Ο τομέας ICT είναι ο τομέας όπου έχει οριστεί η ευρωπαϊκή πολιτική από πλευρά της Κομισιόν. Έχουμε ορίσει ποιες είναι οι κρίσιμες υποδομές έτσι ώστε να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τον εντοπισμό και την αναγνώριση αυτού του είδους ε, των κρίσιμων υποδομών, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια συνεργασία ε, ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και στο κυβερνητικό τομέα και στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει πλήρης ε, συνεργασία στα διάφορα κράτη-μέλη και θα πρέπει να δούμε ποια, ποιος είναι υπεύθυνο γιατί όσον αφορά την ε, ασφάλεια και ποιος μπορεί να ενδυναμώσει την ασφάλειά μας. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση ε, για την συνολική, για τη σφαιρική διαχείριση του κινδύνου. Και η Κομισιόν θα πρέπει να βοηθήσει έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτή η σφαιρική αντιμετώπιση. Τώρα... Σε σχέση με τους πέντε αυτούς τομείς ε, του 2009 δεν θα πω τίποτα, θα περάσω αμέσως στη μελλοντική δράση, διότι πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία στις εξελίξεις που στοχεύουν στην κατεύθυνση που συστήθηκε από τους συντάκτες της έκθεσης που παρουσιάστηκε. Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο πρέπει να θυμόμαστε ότι η ασφάλεια είναι κοινή ευθύνη. Κανείς δεν εξαιρείται από το να υποχρεώνεται να συμμετάσχει σε ένα ρόλο που θα αναλαμβάνει σε αυτή την εικόνα. Αυτό είναι τεράστια σημασία. Γιατί και στο ευρωπαϊκό επίπεδο στη στρατηγική του 2001 σε σχέση με την τελική ρύθμιση εκείνου που πρέπει πρώτος ε, να δρά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι ο τελικός χρήστης είναι ο αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα. Όμως παρόλα αυτά πρέπει να μην αμελήσουμε την ευθύνη κρατών μελών, κυβερνητικών φορέων, ιδιωτικού τομέα επίσης, τομέων, τομεακά, σφαιρικά και συνολικά. Διότι μέσω της τεχνολογίας αυτό συνεπάγεται την εμπλοκή του στην κοινωνία μας. Και έτσι λοιπόν καλούνται τα κράτη-μέλη να δράσουν. Το πιο σημαντικό από όλα σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν ήδη προαναγγεθεί το 2009 στο πρόγραμμα δράσης ε, για την προστασία των υποδομών είναι η ανάπτυξη ενός contingency plan, ενός σχεδίου ετοιμότητας και αντιμετώπισης. Πρέπει να κατανοήσουμε πώς θα συνεργαστούμε από κοινού. Αυτό σημαίνει τι πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο, αποσαφήνιση του τι θα γίνει σε εθνικό επίπεδο και τον επιμερισμό σε σχέση με τα προγράμματα ετοιμότητας που θα πρέπει να συνεισφέρουν και να εμπλέκονται στην ανάγκη για μια ε, συντονισμένη διεθνή δράση. Αυτό έχει τεράστια σημασία διότι όπως είπα ε, στην αρχή το θέμα το ίδιο το οποίο βρίσκεται ε, στη βάση αυτής της συζήτηση είναι το θέμα της διακυβέρνησης, governance. Τα κράτη-μέλη έχουν την πρωτογενή πολιτική ευθύνη πάντα αν κάτι πάει στραβά. Όμως εκείνοι που πρέπει να δράσουν <clears throat> δεν είναι πλέον μόνο κυβερνητικοί φορεί ε, οι εκπρόσωποι. Ο ιδιωτικό τομέα πρέπει να εμπλακεί. Ο ιδιωτικό τομέα πρέπει να κατανοήσει πώ και γιατί και με ποιο κόστο <clears throat> η δράση του θα πρέπει να διαμορφώνεται και να εξετάζεται. Και τελευταίο, εξίσου σημαντικό φυσικά, η συνεργασία. Η συνεργασία διακρατικά μεταξύ των κρατών μελών, με τον ιδιωτικό τομέα, που ήδη <clears throat> θα αποτελεί μια διεθνή πλατφόρμα που θα μπορεί μοχλικά ε, ως μοχλός να δράσει. Αυτό πρέπει να ενορχιστώνεται σε ένα διεθνές περιβάλλον, σε ένα διεθνή περίγυρο. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές και αρχές όσον αφορά την μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και αντοχή του ψηφιακού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Επόμενη διαφάνεια. Η διαδικτυακή ανθεκτικότητα είναι αυτό το οποίο εγγράψαμε στην ημερήσια διάταξη του 2009 ως επίκεντρο δράσεων μεταξύ των κρατών μελών για την άρθρωση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων που πραγματικά θα πρέπει έτσι να προαχθούν σε διεθνές πλαίσιο ώστε να διασφαλίσουμε ότι ενώ θα καλύπτουμε τα θέματα των αναγκών για τη διακυβέρνηση του κυβερνοχώρου θα λαμβάνονται υπόψη τα θεμελιώδη στοιχεία ανοιχτός χαρακτήρας, διαφάνεια, ελευθερία προσπελασιμότητας πρόσβασης. Αυτές οι δραστηριότητες οδήγησαν στην άρθρωση ενός μιας γενικότερης ευρωπαϊκής αρχής για το διαδίκτυο και την ε, ανθεκτικότητα στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω σε σχέση με αυτά τα στοιχεία που αναπτύχθηκαν από κοινού, αναπτύσσονται από κοινού με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο και ήδη αυτό αποτελεί ένα κεκτημένο και ένα προτέρημα, όχι μόνο για την προαγωγή του ευρωπαϊκού επίπεδου μέσω της κοινωνίας ε, των πολιτών και έχουμε και διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών εδώ και κάποιους μήνες, αλλά ακόμα πιο σημαντικό αυτό πρέπει να αποτελέσει προτέρημα για τη συνεργασία μας σε διεθνές επίπεδο. Ο συνάδελφος από την Διπλωματική Εξωτερική Υπηρεσία υπενήχθηκε στην, ε, όσον αφορά την ομάδα εργασίας για την ε, καταπολέμηση του διακυβερνητικού εγκλήματος σε σχέση και με τις δεσμεύσεις και εμπλοκή της Αντιπροέδρου Κρούς και τονίζοντας τις δραστηριότητες όσον αφορά και τις ΗΠΑ για την κυβερνοασφάλεια και όπου συνεργαζόμαστε μέσω των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθεσμικά και με τις ΕΠΑ. Αυτά τα οποία έχουμε εντάξει στο έγγραφό μας που αρθρώνουν τις προτεραιότητες για αυτές τις δράσεις και δραστηριότητες για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και για την κυβερνοασφάλεια σε σχέση με τις, ε, ε, το εγχείρημα που πρέπει να ακολουθηθεί και μέχρι το 2013 αλλά και πιο πρόθεσμα να υπάρξουν ε, ασκήσεις που θα ολοκληρωθούν ετοιμότητας πριν και από το τέλος του 2011 ώστε να μπορέσουμε αυτή την πτυχή του συντονισμού να την θεωρήσουμε ως προτεραιότητα σε σχέση με τα κράτη-μέλη μεταξύ των θεσμικών οργάνων, των διεθνών βήματων, φόρα και φορέων είναι πάρα πολύ σημαντικό από κοινού να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε με αυτές τις πτυχές. Ε, το δεύτερο είναι η ιδιωτική κρατική σύμπραξη. Για τους ίδιους λόγους που ανέφερα πιο πριν. Με την εμπλοκή του ε, ιδιωτικού τομέα δεν μπορούμε να αμελήσουμε την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και πρέπει να αποσταλούν τα σωστά μηνύματα στο εθνικό επίπεδο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ιδιωτική κρατική σύμπραξη, η δημόσια σύμπραξη θα εμπλέκει τους ε, εκπροσώπους ε, ε, με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επένδυση στα θέματα ασφάλειας και να υπάρχει πρόσθετη αξία, όχι μόνο σχετικά αφορά τις επενδύσεις, αλλά προς όφελος της κοινωνίας, κοινωνικό όφελος. Και γι' αυτό οι ιδιωτικές κρατικές συμπράξεις, δημόσιες συμπράξεις είναι στο μέσο που έχει ιδιαίτερο συμφέρον να προαγάγει τη συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ ήδη μπορούμε να προαναγγείλουμε ότι στο εύρο των συζητήσεων με τις ΗΠΑ έχουμε ταυτοποιήσει υλοποιήσει κάποιου τομεί για συνεργασία ο πιθανότερος που θα προαχθεί είναι η εμπλοκή του κρατικού και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των αρνητικών φαινομένων. Πώς θα γίνει αυτό με τη ΣΥΠΑ. Θα γίνει βασιζόμενη και οικοδομώντας στην πείρα και τα, ε, την εμπειρία που έχουμε στα κράτη-μέλη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει προθυμία χωρών όπως Γερμανίας, Ολλανδίας, Σουηδίας, ε, Δανίας ώστε αποκινούμε την εκπόνηση κάποιων στρατηγικών από πλευρά τους να υπάρξει και η εμπλοκή και στον ιδιωτικό τομέα με εταίρους ε, που θα ε, δομήσουν πάνω σε αυτή τη βάση ε, και αμοιβαία με τις ΕΠΑ. Θα έλεγα ότι το ICT δεν είναι μόνο θέμα επικοινωνίας. Υπάρχει εδώ η ε, μεγαλύτερη διάχυση πτυχών του ICT που δίνουν σημασία σε περαιτέρω πτυχές για όλους. Θα πρέπει γι' αυτό να συνεργαστούμε με τις ΕΠΑ για τα θέματα ε, κυβερνοασφάλειας ε, όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, τον επιχειρηματικό τομέα Ωστόσο δεν θα πρέπει μόνο να δούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά δεδομένα ιδιωτών. Πρέπει να δούμε το πώς αμφίδρομα η ροή των στοιχείων και πληροφοριών που διαβιβάζονται πώς σε αυτή την πολλαπλή η ε, διμερή ροή πληροφοριών και στοιχείων πώς όλα αυτά αλλάζουν τη συνολική ας το πω έτσι εικόνα, το σενάριο ε, ε, πραγματών αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αν κάτι πάει στραβά στη Ρουμανία θα έχει επιπτώσεις σε όλο το δίκτυο διαβίβασης ε, πανευρωπαϊκά. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε ότι γεγονότα τα οποία συνέβησαν πριν από κάποια χρόνια στη Γερμανία όπου η εφαρμογή θεμητών μέτρων για την ασφάλεια και για την αντιμετώπιση ενός ενδεχομένου στην εσωτερική αλυσίδα διαβίβασης αμέσως είχε επιπτώσεις λόγω αυτής της ε, διασύνδεσης πανευρωπαϊκά σε άλλες ε, χώρες, σε άλλους εμπλεκόμενους θα έλεγα αρκετές χώρες, ε, Βέλγιο, Γαλλία και άλλες χώρες στην Ευρώπη και για την Ολλανδία τουλάχιστον στην ε, εποχή της κυβερνοασφάλειας ε, μία από τις ε, προτεραιότητες είναι η καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων θα αφήσω τον συνάδελφο να σχολιάσει. Η συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση είναι σημαντικό στοιχείο. Να δούμε πώς θα αρθρώσουμε μηνύματα ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σε σχέση με τις κοινότητες που πρέπει να εμπλακούν και να συνεργαστούν. Και οι διασυνδέσεις, οι οι σύνδεσμοι έχουν και αυτή μεγάλη σημασία. Δεν κάνω λόγο μόνο για τους ISPs, αλλά και για τους παρόχους τεχνολογίας και υπηρεσιών, παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με τους ε, τελικούς ε, χρήστες. Και αναφέρομαι εδώ ιδιαίτερα φυσικά στους χρήστες, στα νοικοκυριά, στους πολίτες, αλλά και πιο σημαντικά λόγω της εμπλοκής στην ε, οικονομική ζωή και στην εμπλοκή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αυτό είναι και αυτό σημαντικό, διότι και αυτό θα βοηθούσε να αρθρωθεί αυτό το οποίο πρέπει να θεωρείται μια νέα απέτηση, νέα πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ενώ οι μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης σε μια διάσκεψη είπαν ότι εδώ όταν εμπλέκονται ε, οι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα και οι ευκαιρίες που προσφέρονται, ευκαιρίες για την προαγωγή των βέλτιστων πρακτικών και προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες αυτές οι δαπάνες από πλευράς ε, κυβερνήσεων και θα πρέπει να δούμε και τον ρόλο των δικτύων και όλα αυτά δεν είναι κάποια επιστημονική φαντασία. Είδαμε πριν από κάποιες ε, εβδομάδες ε, ε, ποιες επιπτώσεις πήρε αυτό το ενδεχόμενο σε σχέση με την πρόσβαση πελατών σε αυτό το δίκτυο. Εν τέλει, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η συνεργασία που θα έχουμε θα υποστηρίζεται πραγματικά από τα κράτη-μέλη. Επόμενη διαφάνεια. Ως αυτό πρέπει να πω πραγματικά ότι η επικοινωνία και η έκβαση των θεμάτων είχαν ήδη συζητηθεί σε ένα άτυπο ε, συνέδριο στο Μπάλατον Φέρετ στην ε, Ουγγαρία ε, τον Απρίλιο, 14-15 Απριλίου 2011 και υπήρξε και μια δήλωση που ήταν η βάση για την άρθρωση συμπερασμάτων, διατύπωση συμπερασμάτων του Συμβουλίου επ' αυτών. Και εδώ μπορείτε να δείτε εν σπέρματι αυτό το οποίο πρέπει να είναι προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή το ένα κράτος να υποστηρίζει αμοιβαία το άλλο. Να υποστηρίζουν αμοιβαία τα κράτη-μέλη σε σχέση με την ε, υιοθέτηση και συμπερασμάτων από πλευρά ε, ε, του Συμβουλίου. Απευθύνθηκε η Επίτροπος κρού ε, στου εκπροσώπους των κρατών μελών ώστε αυτά τα συμπεράσματα του Μπάλατον Φέρετ να ληφθούν υπόψη ώστε να εξοπλιστούν τα κράτη-μέλη και να είναι πρόθυμα τα περισσότερο προηγμένα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν τα λιγότερο εξοπλισμένα και ανεπτυγμένα κράτη-μέλη να αναπτύξουν το δυναμικό τους και αυτό να μπορεί να αντανακλάται σε σχέση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Δεν υπάρχει η ε, ορθή ε, ο, ας το πω έμφαση όπως θα το επιθυμούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για την ενορχίστρωση αυτών των στοιχείων στη μελλοντική πολιτική. Και υπάρχει ήδη έκφραση ενδιαφέροντος που έχει ε, διατυπωθεί από κάποια κράτη-μέλη να υποστηριχθεί αυτή η διεργασία. Ωστόσο από την άλλη πλευρά για να μπορέσουμε να σεβαστούμε τις πρωτογενείς ευθύνες ε, των κρατών μελών των μικρών κρατών μελών, μικρότερων κρατών μελών, πρέπει να υπάρξει διατύπωση αιτήματο αρρωγή και συνδρομή. Και εδώ αυτή η συνεργασία προ αμοιβαία αρρωγή είναι πολύ σημαντική. Και ένα τελευταίο σχόλιο για την ΙΖΑ. Θα έλεγα η συζήτηση για την μελλοντική εντολή είναι πάρα πολύ σημαντική μέσα σε αυτό το πλαίσιο για προτάσεις με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να ενδυναμωθεί η ΙΣΑ πώς θα ενδυναμωθεί, θα ενισχυθεί η συνεργασία και πώς θα υπάρξει ο ορισμός πιο αξιόπιστων ε, στοιχείων και πληροφοριών που πρέπει να αποτελούν τη βάση για την διατύπωση πολιτικών στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο οτιδήποτε μπορεί να <clears throat> αυξήσει τον υφιστάμενο μηχανισμό σε σχέση με το άρθρο 13α της οδηγίας πλαισίου για την ηλεκτρονική επικοινωνία ή σε σχέση με την υποχρέωση υπό το άρθρο 4 Όλα αυτά θα συνεισφέρουν από πλευρά τους ώστε η ΕΝΙΣΑ, η ΕΝΙΣΑ να είναι σε θέση να μπορεί να προβεί σε αξιολόγηση τρίτων εμπλεκομένων ε, για θέματα κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη από που όλοι αναμένουμε θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Thank you. And Mr. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής από την Κομισιόν, παρακαλώ. Είμαστε και με τον συνάδελφο τον Μάρτιν εδώ, ο οποίος θα ξεκινήσει την παρουσίαση και θα καθίσει εκεί για να παραλείψει ορισμένες διαφάνειες ώστε να μην επαναλάβουμε αυτά που έχουν υποθεί από τους προλαλήσαντες. Και μετά εγώ θα σας μιλήσω για την οδηγία σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις. Yes, good morning or good day. Καλή σας ημέρα. Δεν με βλέπετε βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Ε, είχατε πολύ υπομονή και θάρρο. Ε, δεν θα μακρηγορήσουμε εμεί για να μην επαναλάβουμε αυτά τα οποία ήδη έχουν διαμακρών ε, αναφέρει προλαλήσαντε. Γι' αυτό και θα ξεκινήσω με αυτή εδώ τη διαφάνεια. Παραλείποντας προηγούμενες, αλλά θέλει λίγη ώρα αυτό. Ίσως είναι σύμπτωση το ότι υπήρξε επίθεση κατά της Ισπανικής αστυνομίας, κατά του Δουνουτού, κατά του Μιλουσίτη Μπάνκ, που είχε να κάνει με 200.000 ε, δέσμες δεδομένων ε, και αυτά συνέπεσαν με τη δική μας παρουσίαση. Απαντώντας σε μια από εδώ είχε πει ότι Δεν θα πρέπει ούτε από τους στρατιωτικούς ούτε από τον ΝΑΤΟ να περιμένουμε ε, ότι θα αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της κυβερνοασφάλειας. Ο Economist, της προηγούμενου έτους νομίζω, ε, έχει αυτό το εξώφυλλο. Εμείς μιλάμε από την πλευρά της Κομισιόν, δεν, μας, ε, δεν είμαστε αρμόδιοι τόσο για θέματα αμυντικά, όπως γνωρίζετε. Θα σας μιλήσω πιο πολύ για το κυβερνοέγκλημα. Ακούσαμε τους διάφορους όρους αν δείτε και τη μελέτη, σε ό,τι αφορά τα διάφορα cyber, είτε μιλάμε κυβερνοασφάλεια, κυβερνοάμυνα, κυβερνοέγκλημα, το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το να έχουμε μια στρατηγική κυβερνοασφάλεια θα αποτρέψει το κυβερνοέγκλημα. Ίσως όχι είναι η απάντηση. Κατακαιρματισμός επίσης ε, αναφέρθηκε. Είναι και ένα από τα θέματα που θέλουμε και εμείς στην Κομισιόν να αντιμετωπίσουμε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που εμπλέκονται σε ό,τι έχει να κάνει με το κυβερνό. Υπουργεία Εστερικών, Δικαιοσύνης, Αμυνάς, ε, ε, Επικοινωνιών. Ακούσαμε τα περί διεθνών πρωτοβουλειών. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να βγει αν θέλετε από το μικρό του τετραγωνίδιο και να δει την ευρύτερη εικόνα. περνάω και αυτή τη διαφάνεια και πηγαίνω κατευθείαν στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πριν δώσω το λόγο στο συνάδελφό μου, θα ήθελα να αναφέρω ένα πράγμα. Το Συμβούλιο ζήτησε από την Κομισιό να κάνει μια μελέτη σκοπιμότητας ε, για το ε, Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβέρνο Εγκλήματος, κάτι που αναφέρεται και στην εσωτερική στρατηγική ασφάλειας. Μερομηνία είναι το 2013, να είναι επιχειρησιακό τότε το κέντρο αυτό. Πολύ πρόσφατα λοιπόν ξεκίνησε η μελέτη σκοπιμότητας με θέμα ένα τέτοιο κέντρο τίποτε το πρέπει να κάνει. Θα το απαντήσει η μελέτη σκοπιμότητας και θα μας πει και το πού θα έχει την έδρα του. Μια πρώτη, ένα προσχέδιο το περιμένουμε στα τέλη του έτους και την έκθεση ελπίζουμε να την έχουμε στις αρχές του 2012. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα για να ε, ξεκινήσει και να κάνει και τις πρώτες του, να αναλάβει τις πρώτες του εργασίες στο κέντρο αυτό. Εδώ έχετε γραφικά έτσι την ε, λειτουργία του κέντρου τι σημαίνει ουσιαστικά αυτό το κέντρο. Το κέντρο αυτό υποτίθεται ότι θα συνενώνει κάποια κομμάτια του παζλ. Κατάρτιση και ε, επικοινωνία και μετάδοση των γνώσεων που είναι μια συνιστόσα. Επίσης, η σημαντική ενημέρωση ότι γίνεται ένα κυβερνό έγκλημα πρέπει να εντοπιστεί, να επισημανθεί, μετά η έκθεση να περάσει σε μια εθνική πλατφόρμα συναγερμού, μετά να γίνει αξιολόγηση της πληροφορίας και αν θεωρηθεί σκόπιμο τα δεδομένα αυτά θα μεταφερθούν στο, στην πλατφόρμα του κέντρου κυβερνοεγκλήματος που θα αναλυθούν, θα εμπλουτιστούν θα γίνουν δηλαδή επιχειρησιακή πληροφορία, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για λόγους εκπαίδευση, κατάρτιση κτλ. Ελπίζουμε, όπως καταλαβαίνετε, από αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος να μπορούν να ξεκινούν και κάποιες έρευνες. Κίνδυνοι. Αυτό το κέντρο σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει και καλύπτεται αυτό και στη μελέτη της θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα του ορισμού αυτής της διαπαφής μεταξύ κυβερνοεγκλήματος και κυβερνοασφάλειας ευρυτέρα τη ενία. Δεν ακούσαμε βέβαια πολλά για το, λόγο, για το ρόλο των κρατών μελών, αλλά σίγουρα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τι των κρατών μελών. Γιατί η αρχή είναι πολύ απλή. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση από τα κράτη-μέλη που να μεταφέρεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα πρόβλημα που το βλέπουμε καθημερινά ε, και στη Europol. Έχει να κάνει λέει, με οποιαδήποτε άλλη μορφή εγκλήματος. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία, δεν υπάρχει καμιά προσθέμενη αξία. Επίσης, υπάρχει ήδη ένα μεγάλο ε, αριθμός καθηκόντων που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Η μελέτη σκοπιμότητας θα πρέπει να, ασκήσει, να ε, εκτιμήσει με κριτικό πνεύμα το εφικτό ε, όλων αυτών των καθηκόντων. Ο συνάδελφός μου τώρα θα σας μιλήσει για την νομική πρόταση που θα διατυπωθεί σύντομα και θα σας μιλήσει και για την ομάδα εργασίας με τη turn it off. turn it off The Thanks very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσθέσω και εγώ την παρέμβασή μου δίνοντας περαιτέρω επεξηγήσεις ε, για αυτή την ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου που διοργανώθηκε, θεσπίστηκε σε υψηλό επίπεδο ε, υπαλλήλων. Έχει το, την κυβερνοδιαχείριση και το κυβερνοέγκλημα ο συνιστώσεις. Για το κυβερνοέγκλημα συμφωνήσαμε σε τρεις προτεραιότητες σε επίπεδο εργασίας. Η δια διαχειρισιμότητα ε, αμοιβαία και πρέπει περισσότερο να γίνουν, περισσότερα να γίνουν στο επίπεδο διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το θέμα κατάχρησης ε, και των ε, πρωτοκόλων ή των πηγών τραπεζών δεδομένων διευθύνσεων και ονομάτων και σε σχέση και με τα ονόματα και κώδικες σε σχέση με το διαδίκτυο και μητρώα και όσον αφορά τα θέματα διαδικτύου είναι πάρα πολύ περίπλοκη αυτή η διαδικασία διαδικασία αλλά πρέπει να καλυφθεί και να αντιμετωπιστεί. Είναι μία από τι προτεραιοτητε αυτη τη ομαδα εργασια λοιπόν αυτή. Οι αλλε δύο προτεραιότητες είναι η καταπολέμηση τη παιδικής πορνογραφίας. Θα έχουμε μία συνάντηση στι 28-29 Ιουνίου σε σχέση με αυτό το θέμα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας σας έχουμε και εκπροσώπους επαΐοντες ε, των κρατών μελών που θα συμμετάσχουν θα αντιμετωπίσουν προτάσεις από πλευράς τεχνολογίας για την απάλληψη διαγραφή εικόνων παιδικής πορνογραφίας από το διαδίκτυο καθώς επίσης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων την σχέση, σε σχέση με τον συσχετισμό με σχέση με τηλέφωνα άμεσης ε, δράσης ε, και δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης ε, και σε σχέση και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τη Σύμβαση για την καταπολέμηση του Κεβερνού εχουμε έχουμε νέα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα κυρώσει αυτή τη σύμβαση. Έχουν υπογράψει όλα τα κράτη-μέλη αλλά εννέα δεν έχουν ακόμα κυρώσει αυτή τη σύμβαση και συχνά τονίζεται από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εμπλεκομένους ότι πρέπει να θέσουμε εντάξει τα του οίκου μας πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτού προτείνουμε σε κράτη-μέλη που δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσχωρήσουν και να κυρώσουν αυτή τη σύμβαση. Κοινή προσπάθεια από πλευρά τη Σεσίλια Μάνστρομ Επιτρόπου και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τις εννέα κράτη, ε, χώρες μέλη που δεν έχουν ακόμα προσυπογράψει, ε, δεν έχουν επικυρώσει ακόμα αυτή την σύμβαση. Αυτή είναι μια κοινή δράση όσον αφορά αυτή τη Τώρα, συνιστόσα του ε, ποινικού ε, κώδικα για την αντιμετώπιση εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο έχουμε αν ήδη καλύψει το θέμα της, ε, αναφερθεί στο θέμα της ανθεκτικότητας ή αντοχής ε, των υποδομών, την ε, συνιστόσα επίσης σε σχέση με διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις, αλλά και από πλευράς ποινικού δικαίου, ποινικού κώδικα προσπάθειες αντιμετώπισης αυτής της, αυτού του φαινομένου. Από το 2005 έχουμε μία απόφαση πλαίσιο όσον αφορά την, τις δράσεις στα δίκτυα πληροφορικής και πληροφορίας πάνω κάτω 20 κράτη-μέλη από τα 27 κράτη-μέλη έχουν υλοποιήσει αυτές τις ε, διατάξεις, αυτές τις προδιαγραφές. Έχουμε επίσης και το ε, δεδομένο του πλήγματος ε, στην Εστονία, της επίθεσης στην Εστονία που αφύπνισε πάρα πολλούς από εμάς τα προβλήματα και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνειδητοποίησαμε ότι οι επιθέσεις μεγάλης κλίμακας είναι πλέον κάτι συνηθισμένο και έχουν πολύ μεγάλες, παίρνουν πολύ μεγάλες διαστάσεις και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν, να καταπολεμηθούν από εμάς. Και τώρα κατεύθυνση προς τη νέα πρόταση που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2010 με τη νέα οδηγία σε σχέση με επιθέσεις στα συστήματα πληροφορικής βασίζονται ακριβώς τα στοιχεία σε αυτή την ανάλυση αυτής της απειλής και το ότι πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε επιθέσεις μεγάλης κλίμακας. Γίνεται ε, αναφορά επίσης στα ε, δίκτυα bot, bots που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ε, δίκτυα ε, οικονομικών εγκεφάλων που εμπλέκονται σε μια τέτοια επίθεση ταυτόχρονα και μπορούν να οδηγήσουν στην κατάρρευση ολόκληρων συστημάτων. Αναφέρομαι εν συντομία σε αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναφέρομαι στα κυριότερα καινοτόμα στοιχεία. Ίσως όπως γνωρίζετε το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων και δικαιοσύνη. την προηγούμενη Παρασκευή υιοθέτησε μια γενική ε, κατεύθυνση, ένα γενικό προσανατολισμό επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γενικά θα σχολιάσω και αυτή την γενική η προσέγγιση από πλευρά του Συμβουλίου. Στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Επιτροπή ΛΥΜΕ, που είναι το κύριο κοινοβουλευτικό όργανο στην Ευρωβουλή για τη συζήτηση αυτών των θεμάτων, έχουν ήδη συζητήσει δύο ή τρει φορέ αυτά τα θέματα και θα υπάρξει και μια κρόαση από αυτών των θεμάτων και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να ε, τους κάνουμε να συμμετάσχουν σε αυτά τα τεκτενόμενα. Υφίστανται κυρώσεις λοιπόν οι, χρήση, οι αυτών των εργαλείων των μέσων, τα αποκαλούμε μέσα η εργαλεία εργαλεία, tools, διότι δεν θέλουμε να εξειδικεύσουμε περισσότερο τέτοιου είδους ε, μεγαλύτερες επιθέσεις ε, μέσω άλλων. Ε, χρησιμοποιούμε τον όρο γενικά tools. Επιβάλλονται κυρώσει σε σχέση με τη χρήση αυτών των tools, μέσων ή εργαλείων και των χρηστών για παράνομη πρόσβαση, παράνομη παρενόχληση, παρεμπόδιση, παρακόλληση και η illegal interception, η παράνομη εκμετάλλευση, ε, η σύλληψη στοιχείων είναι κάτι το οποίο ως νέο στοιχείο εμπεριέχεται σε αυτή την απόφαση πλαίσιο σε σχέση με την πρότασή μας ε, βελτιώνεται η, συνεργασία των αστυνομικών οργάνων και η επιβολή του νόμου βελτιώνοντας ε, τους συνδέσμους ε, όσον αφορά τα σημεία που είναι σύνδεσμοι έχουμε επίσης και συγκεκριμένη περίοδο ετοιμότητας που προβλέπεται εκείνο το οποίο υπήρχε στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο κείμενο έχουμε ένα νέο στοιχείο την οκτάωρη αυτή περίοδο για την εξέταση κατεπιουσών αιτήσεων από τα κράτη-μέλη σε περίπτωση ε, κυβερνοεπιθέσεων ως σημαντικών υποθέσεων και των αναγκαίων αντιδράσεων ως ένδειξη ότι θα υπάρξει συμμετοχή σε αυτή την αντίδραση. Σημαντικό να συμπεριλαμβάνεται αυτό. Διαβουλευόμενοι αυτού είπαμε ότι είναι εφικτό το πλαίσιο της ε, οκτάωρης αυτής ετοιμότητα. Προθυμία και ετοιμότητα συλλογή στατιστικών στοιχείων ε, για τέτοιου είδου κυβερνοεγκλήματα, κυβερνοεπιθέσει, ε, cyber attacks που ήταν μάλλον εμβαλωματικού χαρακτήρα μέχρι σήμερα. Και τέλος εξίσου σημαντικό, αυξάνεται το επίπεδο των κυρώσεων σε μέγιστη φυλάκιση διαιτή τους διάρκειας καθώς επίσης και σε ιδιαίτερα ε, σοβαρές περιπτώσεις σε περίοδο πενταετούς ε, φυλάκισης. Προηγούμενα υπήρχε ε, ως βασική κύρωση η φυλάκιση ενός έτους και πρέπει νομίζω αξίζει να τονιστεί ότι πρόκειται για μέγιστες ποινές που εξετάζονται υπό το πρίσμα του ποινικού δικαίου θα είναι ελάχιστες αυτές οι ποινές αλλά εμείς αυξάνουμε το επίπεδο φυλάκισης ε, σε ένα μέγιστο ε, ε, επίπεδο. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τα ελάχιστα επίπεδα σε ένα μέγιστο όριο. Θέλουμε λοιπόν εκείνα τα κράτη-μέλη που έχουν τριετή περίοδο, προβλέπουν τριετή περίοδο φυλάκισης να την αυξήσουν σε πενταετή. Και αυτό σε σχέση με ε, τις δεδομένες αυτές παραβάσεις. Προσπαθούμε να αυξήσουμε τα ε, μάξιμα, τις ε, μέγιστες ποινές, λέγοντας τα κράτη-μέλη είναι πολύ σοβαρά δικήματα αυτά και πρέπει με σοβαρό τρόπο να τιμωρούνται. Έχουμε τρεις επιβαρυντικές ε, περιπτώσεις ως συνιστώσεις όταν υπάρχει υποτροπιασμός πολλαπλά με τέσσερα ας πούμε αδικήματα ή τέσσερις επιθέσεις το νέο είναι η χρήση ενός συγκεκριμένου botnet, ενός tool, εργαλείου για την πρόκληση σημαντικής ε, ζημιάς ε, ή ε, εμπλοκής τέτοιων εργαλείων. Το επόμενο στοιχείο είναι όταν χρησιμοποιείται το spoofing για μια τέτοια επίθεση ή θα μπορούσε κανείς να το αναφέρει ως χρήση ε, υποκλαπής ταυτότητας για την άσκηση αυτής της επίθεσης. Βλέπουμε εδώ και μια ιδιαίτερα επικίνδυνη συνιστόσα. Εκμετάλλευση της ανθρώπινης της εμπιστοσύνης ε, χρηστών του διαδικτύου όταν αποστέλλεται μια πλασματική ταυτότητα ε, συνδιαλεγωμένου με κάποιον ο οποίος την έχει υποκλέψει αυτήν. Και βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηρή σε σχέση με αυτό. Υπάρχουν διαφορετικές λεπτομέρειες σε σχέση με τα στοιχεία που αποστέλλονται με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. Πολλοί δεν το προσέχουν αυτό. Μπορεί να φαίνεται ως ε, πραγματικό άτομο μιας ε, ε, οργάνωσης κάποιος και βλέπουμε ότι εδώ μπορεί να υπάρχει το ενδεχόμενο ιού που μπορεί να διαδοθεί και να μολύνει δίκτυα μέσω, όλοκληρο μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και αυτό μπορεί να, με τη διάχυση που θα έχει να βλάψει ολόκληρα δίκτυα. Έχουμε ακούσει από αρκετούς επαΐοντες ότι υπάρχουν επίσης περιπτώσεις ε, τέτοιων ε, επιθέσεων κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, χρησιμοποιώντας η επιτιθέμενοι πλασματικά την ταυτότητα κάποιου επιτρόπου ώστε να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνη με τους υπαλλήλους της Επιτροπής και να ασκηθεί αυτή η επίθεση. Θέλουμε λοιπόν αυτή την πτυχή της υποκλοπής προσωπικότητας να την αντιμετωπίσουμε. Την προηγούμενη Παρασκευή όπως είπα μια γενική, ένας γενικός προσανατολισμός υιοθετήθηκε από το Συμβουλίο. Καλοχαιρετίζουμε, δεχόμαστε ε, με ιδιαίτερη ιδιαίτερη ευχαρίστηση στην πρόθεση της Ουγγρικής κυβέρνησης ε, που προεδρεύει στο Συμβούλιο να προαγάγει αυτά τα θέματα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένας συμβιβασμός αυτός που επετεύχθη. Δεν είναι η αρχική πρόταση που είχε διατυπωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενώ ταυτόχρονα εκτιμούμε πάρα πολύ τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν έχουμε ξεχωριστή άποψη για αρκετούς συμβιβασμούς που εμπεριέχονται στο, κείμενο με συγχωρείτε. και εντάχει θα αναφερθώ σε αυτές τις πτυχές γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε σε σχέση με αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν οι παναχωρήσεις σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αρχίζω με τα θετικά. Καλωσορίζει Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αύξηση των επιπέδων των κυρώσεων σε ένα μέγιστο δύο ετών από το προηγούμενο επίπεδο ενός έτους ε, ποινών καλοχαιρετίζει το σθένος να αντιμετωπιστούν τα, οι περιπτώσεις κυβερνοεγκλημάτων με στεναρότητα, με σθένος. Νέες επιβαρυντικές προτάσεις ε, ως στοιχεία προστίθενται σε αυτή την πρόταση και υπάρχει ένα τέτοιο επιβαρυντικό στοιχείο όταν γίνονται αυτά, αυτές οι επιθέσεις εναντίον ενός κέντρου κέρια σημασία υποδομών. Εκεί η προτινόμενη ποινή είναι 5 ετών. Επίσης εκτιμούμε την ανάγκη ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υπάρξει η τιμωρία σε σχέση με συγκεκριμένη χρήση εργαλείων στις κυβερνοεπιθέσεις. Πρέπει να ενισχυθεί επίσης να ενδυναμωθεί η συνεργασία κρατών μελών ε, σε σχέση με την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και πρέπει να Υπάρχουν και στατιστικά στοιχεία σε σχέση με όλα αυτά. Όλα αυτά είναι θετικά στοιχεία σε σχέση με τη γενική προσέγγιση αυτών των θεμάτων από το Συμβούλιο. Τώρα, λιγότερο θετικά είναι τα στοιχεία που αφορούν την έκβαση σε σχέση με την εφαρμογή των επιβαρυντικών στοιχείων που μειώθηκε, σε, συρρυκνώθηκε σε δύο μόνο ε, περιπτώσεις παραβάσεων. Τα άρθρα 4 και 5 εμπλοκή και παρεμβολή σε σχέση με παράνομες δράσεις όσον αφορά συλλογή στοιχείων και τα άλλα δύο για το άρθρο 3 και 6 για την παράνομη πρόσβαση και την παράνομη ε, συλλογή. Εκφράζουμε τη θλίψη μας για αυτό το γεγονός διότι ε, το έβρος της οδηγίας βασίζεται στην γνώση, στην συλλογή και υφή περιπτώσεων που δεν είναι ίσονος σημασίας. Όλες αυτές ε, οι περιπτώσεις δεν είναι ίσονος σημασία θέματα. Και η ανησυχία μας είναι ως κύριο μέλημα αυτό. Δεν θέλουμε φυσικά να υπάρξει υπερβολική ποινική κύρωση όσον αφορά ίσονος σημασίας ε, ε, παραπτώσεις παραβιάσεις ή παραπτώματα σε σχέση με νέους ε, που διαπράττουν κάποια αδικήματα. Θέλουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο σε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις και στη συνιστόσα του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης, Κλειβόμαστε ε, για το ότι δεν μας υποστήριξε το Συμβούλιο στην διασφάλιση του άρθρου 99 5 όσον αφορά την επιβαρημένη χρήση ε, υποκλοπής ε, στοιχείων προσωπικότητας κάποιου ε, άλλου ατόμου. Επεξηγήσαμε προς το Συμβούλιο ότι αυτό γίνεται όλο και πιο συχνά σε σχέση με κυβερνοεπιθέσεις. Ολοκληρώστε παρακαλώ γιατί δεν υπάρχει επαρκής χρόνος σε σχέση με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με πλασματική πλασματική ταυτότητα. Το επιχείρημα από πλευρά Συμβουλίου ήταν ότι πρέπει να υπάρχει ένα γενικό μέσο για την καταπολέμηση της ε, πλασματικής χρήσης ταυτότητας. Όμως εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο αυτό το αδίκημα. Είναι όλο και πιο συχνές ε, οι περιπτώσεις ε, που κάνουν χρήση οι εγκληματίες αυτής της μεθόδου. Επίσης, σε σχέση χειραγώγησης μέσων για την ε, τελική ε, έκβαση σε χρήση πολλαπλών τέτοιων ε, εργαλείων αυτό δεν θεωρήθηκε επιβαρυντική περίπτωση άσχετα από τις επιπτώσεις της επίθεσης. Η δική μας πρόταση είχε αρκετές εγγυήσεις που τη συνόδευαν ότι σε περιπτώσεις μη ε, σε περιπτώσεις σημαντικών επιπτώσεων θα υπήρχε αυστηρή εφαρμογή του νόμου και αυστηρή ποινή σε σχέση με την ε, δυνατότητα να μπορούν να αποτρέπονται ε, πολλοί από τέτοιου είδους πράξεις όμως βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η ενδεχόμενη απειλή και όμως δεν αντιμετωπίστηκε όπως προτείναμε εμείς σε συζητήσεις σε σχέση με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ, που έχουν γίνει μέχρι σήμερα επ' αυτού του θέματος, πρόκειται για κυβερνοεπιθέσεις. Δεν επιλύονται οι, ε, συνολικά οι, όλες οι πτυχές των, του κυβερνοεγκλήματος επικεντρωνόμενοι σε αυτή την πτυχή ε, για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος χρειάζονται και άλλοι, άλλα μέτρα τα οποία πρέπει να ε, συνοδεύουν μια τέτοια πρόταση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκάλερ για ένα τελευταίο ερώτημα. Ναι, ευχαριστώ. Δεν μπορώ να θέσω κάποιο θέμα ε, ειδικό και ουσίας, αλλά το συμπέρασμα που συνάγω εγώ από, αυτό, από αυτή την ακρόαση είναι ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αντιληφθεί τα προβλήματα με χαρά άκουσα ότι από ό,τι φαίνεται στις 6 Ιουνίου έγινε αυτή η διεπηρεσιακή συνάντηση σε επίπεδο γενικών διευθυντών στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Βιλαλόγκα. Και σε ό,τι αφορά την ΕΙΕΔ ήταν ο Ποπόφσκι ο αναπληρωτής ε, γενικός ε, διευθυντής. Αυτό είναι γενικός δραματέας. Ε, Αυτό πολύ θετική εξέλιξη. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς τον κύριο Βιλαλόγκα. Σε ποιο επίπεδο στην ΕΙΕΔ θα γίνει περαιτέρω επεξεργασία του, θα φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να είναι καθημερινή εργασία του κυρίου Ποπόφσκι αυτή. Και από ό,τι είδα, τη δική σας ιδιότητα ε, είναι κάπως γενικότερη. Υπάρχει μια μονάδα συγκεκριμένη, υπάρχει ένα σημείο εστιακό επαφή συγκεκριμένο στην ΕΕΔ και σε ό,τι αφορά το κέντρο ε, του εγκλήματος και τη μελέτη σκοπιμότητας και για το θέμα της έδρας. Είναι σχεδόν διπλάσιες οι δομές που έχουμε και ίσως υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ ΕΕΔ και Κομισιόν. Πού θα μπορούσε να έχει την έδρα του αυτός ο νέος οργανισμός, κάπου στο ενδιάμεσο, κάπου στο μεσοδιάστημα. Να δούμε λοιπόν τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Yes, uh, very quickly, as I mentioned before, there are, there are several... Όπως προείπα, υπάρχουν στην, εξωτερική, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης διάφορες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με θέματα ασφάλισης. Έχουμε τον κύριο Ρίτς Ράιτ ε, που ασχολείται με τα θέματα της πρόληψης και της πολιτικής Έχουμε λέξη ε, κάποια εμπειρογνωμοσύνη και μάλιστα θα προσλάβουμε και άλλους εμπειρογνώμονες. Επειδή αυτή, αυτό το θέμα προσλαμβάνει σημασία. Εγώ τελώ χρέη ε, διευθυντή αυτής της μονάδας που ε, σύντομα θα ε, ε, καλυφθεί μάλλον μέσα στο καλοκαίρι γιατί θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω, λέει ο όλους τους ομιλητές και να κηρύξω το τέλος της συνεδρίασης.